Colleagues, uh, please take your seats and we can uh, begin. Συναδέλφοι, καλημέρα σας. Συναδέλφοι, παρακαλώ καθίστε. I'm uh, for those colleagues from SEDE, I'm ε, για τους συναδέλφους της ΕΝΤΑ, εγώ είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και φυσικά η κυρία Φωτήγα είναι ε, πρόεδρος της Επιτροπής ΕΝΤΑ και από κοινού και με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στην ε, ακρόαση για την ε, διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκληση για την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια. Η συνάντηση αυτή ετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Πολλοί κόσμος ήθελε να γίνει μια κοινή συνεδρίαση μεταξύ των επιτροπών μας και η κυρία Φορτίγα μου το είχε αναφέρει ξανά στο παρελθόν και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι εδώ στην αίθουσα ε, είναι πολύ σημαντικό που συναντώνται για να συζητήσουν για αυτά τα συνοριακά ζητήματα. Χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους βρέθηκε χρόνος για να συναντηθούν από κοινό αυτές οι επιτροπές και να συζητήσουν τα τόσο ευαίσθητα ζητήματα της διαχείρισης των συνόρων. Σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι που βρήκατε χρόνο και καταφέραμε να συναντηθούμε εδώ. Πώς θα οργανώσουμε τις εργασίες μας. Ε, πρέπει να πω ότι με τις δύο επιτροπές μαζί δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους με τόσους τίτλους σε ένα τόσο μικρό χώρο. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί για να μην κάνουμε λάθη. Λοιπόν, εγώ προσφέρθηκα εθελοντικά για να προεδρεύσω το πρώτο πάνελ, αλλά θα παρουσιάσει ο καθένας τους δικούς του ομιλητές, σωστά, κυρία Πρόεδρε. Είναι περίπλοκο, αλλά θα το καταφέρουμε. Εγώ θα παρουσιάσω λοιπόν τους ομιλητές που σχετίζονται με τη ΛΥΜΠΑ και η κυρία θα παρουσιάσει τους ομιλητές που σχετίζονται με την ΣΕΝΤΕ. Ωραία λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο για να ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε το πρώτο πάνελ. Θα θέλατε να παρουσιάσετε τους ομιλητές σας για αυτό το πάνελ. Καλησπέρα για άλλη μια φορά κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σας ε, υποδέχομαι σε αυτή την εξαιρετική συνάντηση με πολλές προσωπικότητες και θέλουμε όλοι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Έλερ για την ε, πρωτοβουλία του. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω παρουσιάζοντας τους εξαίρετους ε, ομιλητές του πρώτου πάνελ τους οποίους υπέδειξε η Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Επειδή το θέμα αφορά τους συνοριακούς ελέγχους και την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των οργανισμών και των διεθνών οργανισμών αποφασίσαμε να ακούσετε τις απόψεις ορισμένων ε, ε, πολύ σημαντικών, κρίσιμη σημασία οργανισμών. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας προσθέσω για άλλη μια φορά ουσιαστικά τον υπονάβαρχο Ενρίκο Κρεντεντίνο ο οποίος είναι διοικητής ε, της UNAFOR Sofia διοικητής δηλαδή της αποστολής που ακόμα ε, ε, δεν έχει λήξει, βρίσκεται στη δεύτερη φάση της, στο πρώτο κομμάτι της δεύτερης φάσης των επιχειρήσεων, στη Μεσόγειο θάλασσα, διασώζοντας ε, πρόσφυγες δημιουργήθηκε αυτή η επιχείρηση γιατί μας απασχόλησαν, απασχόλησε το δράμα που συντελείται στην Πεσόγειο και έτσι αποφασίσαμε να στείλουμε μια ναυτική αποστολή τη δεύτερη και ελπίζουμε να είναι το ίδιο επιτυχής με την Αταλάντα. Ο υποναύρχος κ. Πιεντεντίνο έχει ξαναβρεθεί σε συνάντηση της ΕΝΤΕ και τότε σας παρουσίασε στις επιχειρήσεις της Uniformat και τώρα θα μας παρουσιάσει τις περαιτέρω εξελίξεις των γεγονότων. Να σας παρουσιάσω επίσης τον, την πρέσβυρα Φραντσέσκα Ταρντιόλη η οποία είναι αναπληρώτρια ε, βοηθός γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ αρμόδια για επιχειρήσεις. Μετά από την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ για την κίνηση των ε, επιχειρήσεων στο Αιγαίο. Είναι πολύ σημαντική και η δική της άποψη. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, ας ακούσουμε τα μέλη του πάνελ και δίνω το λόγο στον συνάδελφο μου τον κύριο Μωράης για να μας παρουσιάσει του δικά του μέλη του πάνελ. Ευχαριστώ πολύ Άννα. Έχω δύο μέλη στο πάνελ, τον κύριο Φαμπρίς Λετζέρη εκτελεστικό διευθυντή της Frontex και για τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ αλλά και της ΣΕΝΤ δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση Frontex ξεκίνησε από έναν οργανισμό με ένα σύνολο στόχων σε έναν οργανισμό που επεκτάθηκε ε, πάρα πολύ και αυτό θα είναι και το αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα. Ο κ. Λετζέρη είναι εξαιρετικά πολύ άσχολο οπότε τον ευχαριστούμε που βρίσκεται μαζί μα σήμερα. Δεύτερο μέλο ο κ. Όντριτ Μαρτινού, αναπληρωτή διευθυντή τη Ευρωπόλ και πάλι εδώ έχουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό ο οποίο έχει επεκτείνει τι δραστηριότητε του ζωτική σημασία για τι σημερινέ μα συζητήσει. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που βρίσκεται μαζί μα σήμερα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια παρουσίαση για τους συναδέλφους που μόλις μπήκαν στην αίθουσα η ΛΥΜΠΕ και η ΣΕΝΤΕ συνεδριάζουν μαζί σήμερα διότι μετά από μια πρόταση του Christian πριν από μερικούς ε, μήνες ε, η κατάσταση στα σύνορα έχει γίνει πιο περίπλοκο ε, ζήτημα οπότε η συνεργασία μεταξύ Frontex, Europol, Eurojust, Unifor και άλλων οργανισμών αποτελεί πλέον πραγματικά, αλλά πολύ περίπλο, πραγματικότητα, αλλά πολύ περίπλοκη πραγματικότητα. Δεν αφορά μόνο τη λαθρεία διακίνηση και το λαθρεμπόριο. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπως ε, το θέμα των σύνοριοφυλακών. Οπότε είναι πήγοντα τα ζητήματα αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργούν αυτές οι, αυτοί οι οργανισμοί και πώς συνεργάζονται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση για το πώς οι επιμέρους οργανισμοί βλέπουν το ρόλο τους και ο πρώτος ομιλητής είναι ο υπονάβροχος Ενρίκο Κρεντεντίνο, ο οποίος θα πάρει πρώτος λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να βρίσκομαι εδώ μαζί με τους συναδέρφους από την Frontex, τη Europol, τη Eurojust. Όλοι αποτελούμε μέρος ε, της ε, γενικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είναι σημαντικό όμως να συνεργαζόμαστε και με το ΝΑΤΟ, διότι παρότι λειτουργούμε σε διάφορες περιοχές, μοιραζόμαστε την ίδια περιοχή, τη Μεσόγειο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλοι μαζί να συζητούμε αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Uniform Med, λοιπόν, πριν ένα χρόνο, 16 ναυτικά μίλια από την ε, ακτή της Λιβύης, βόρεια της Τρίπολης, ε, ε, πέθαναν 10 μετανάστες και αυτό ήταν το χειρότερο ατύχημα. Δύο αργότερα, στις 13 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε Συμβούλιο Εξωτερικών και υιοθετήθηκε ένα σχέδιο και το ε, UNOFARMED ήταν το δεύτερο θέμα στη μερίσια διάταξη. Έχουμε λοιπόν πολύ σύντομο χρονικό διάγραμμα. Πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε τους ε, διακινητές ανθρώπων ε, ώστε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του προβλήματος. Η αναζήτηση και διάσωση δεν αποτελεί μέρος της εντολής, αλλά η διάσωση ανθρώπων αποτελεί διεθνή υποχρέωση. Εμείς οι ναυτικοί ποτέ δεν αφήνουμε κάποιον ε, σε κίνδυνο στη θάλασσα. Στη θάλασσα υπάρχει μόνο ένας νόμος, όποιος βρίσκεται σε κίνδυνο θα πρέπει να διασωθεί. Έχουμε σώσει λοιπόν πάνω από 12.000 ανθρώπους ε, σήμερα. Τα δεδομένα που βλέπετε εδώ μας τα έχει δώσει η Frontex, ε, είναι αφορούν το 2015 και σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέφτασαν στην Ευρώπη, το 82% μέσω της Ανατολικής Οδού, μέσω των Βαλκανίων, ενώ το 16% επέλεξαν το δρόμο της ε, Κεντρικής Μεσογείου. Πέρσι ε, υπήρχε ε, ίση κατανομή ανάμεσα στην Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για διάφορους λόγους είχαμε μεταφορά των ρευμάτων στο δεύτερο εξάμεινο. Ένας από τους λόγους ήταν ότι η Αίγυπτος ε, ε, ελέγξε πιο αποτελεσματικά τα σύνορά της. Ήταν λοιπόν πιο δύσκολο να περάσει κανείς ε, στη Λιβύη. Επίσης, ο, η νότια διαδρομή είναι η πιο επικίνδυνη. Τους περισσότερους θανάτους τους είχαμε εντός των εδαφικών υδάτων της Λιβύης και Η Frontex ε, κινητοποιήθηκε στις ακτές ε, της Λιβύης ε, και έτσι απέτρεψε αρκετούς διακινητές. Το 2016 η κατάσταση παραμένει σχεδόν όμοια. Το 88% επιλέγει την Ανατολική Οδό, το 18% την Νότια Οδό, αλλά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μετά το κλείσιμο των Βαλκανίων έχουν αλλάξει τα πράγματα και βλέπουμε αντιστροφή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Το 55% ήρθαν από τον Νότο, ενώ το 45% από τα Ανατολικά. Έχουμε δει λοιπόν αλλαγή. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να αξιολογήσουμε αν το κλείσιμο των Βαλκανίων θα ε, επηρεάσει την ε, κατάσταση, αλλά νομίζω πως ναι. οι μετανάστες που δεν θα μπορέσουν να έρθουν από τη Στεριά θα προσπαθήσουν να έρθουν ε, κατευθείαν από τη θάλασσα στην Ιταλία, από την Τουρκία, το Λίβανο, τη Συρία, ε, την Αίγυπτο ή μέσω του Σουδάν στη Λιβύη. Αυξάνονται λοιπόν τώρα οι μεταναστευτικές ροές και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση το καλοκαίρι. Εδώ βλέπετε την περιοχή της Αιγίου ε, η γαλάζια περιοχή είναι αρκετά μεγάλη και δραστηριοποιούμεθα από τα σύνορα της Τινησίας ε, προς τα βόρεια και είναι περιοχή πολλών επιχειρήσεων. Έχουμε την Τρίτον, έχουμε τη ε, Frontex, την επιχείρηση Ποσειδών με τον ΝΑΤΟ και κάποιες ανεξάρτητες ε, επιχειρήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχουμε λοιπόν πολλά σκάφη, πολλούς ανθρώπους ε, που ε, λειτουργούν με πολύ καλό συντονισμό. Επίσης έχουμε πολύ καλό καταμερισμό των καθηκόντων μας με το ΝΑΤΟ. Επικεντρωνόμαστε κυρίως έξω από τα εδαφικά ύδατα της Λιβύης. όπου πραγματοποιούνται πάνω από το 90% των ε, επιχειρήσεων διάσωσης. Επίσης, οι ροές από την Αίγυπτο σταμάτησαν πέρσι τον Νοέμβριο, αλλά ξαναξεκίνησαν μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Έξι μεγάλα αλλιευτικά σκάφη είδαμε από την Αίγυπτο προς την Ιταλία μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο. Και αυτό συνδέεται μάλλον με το κλείσιμο ε, της οδού των Βαλκανίων. Σήμερα λοιπόν ε, έχουμε κινητοποιηθεί σε διεθνή ύδατα, μας έχει επιτραπεί αυτό. Έχουμε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και προτού προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, στις 2 Οκτωβρίου, πολύ συχνά οι διακινητές προσπαθούσαν να συνοδεύσουν ε, τα ε, σκάφη μέχρι τα διεθνή ύδατα και προσπαθούσαν ε, έτσι ε, να πετύχουν διάσωση και να ε, ε, ξαναπάρουν τα σκάφη και να τα επιστρέψουν στη Λιβύη. Από τις 2 Οκτωβρίου όμως πια οι διακινητές δεν έχουν ελεύθερο περιθώριο ευελιξίας στα διεθνή ύδατα, διότι θα συλληφθούν από εμά. Έχουν χάσει λοιπόν όλα τα ξύλινα και φουσκωτά σκάφη τους. και έτσι δεν μπορούν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν μετά τις επιχειρήσεις διάσωσης. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και περιμένουμε τώρα να δημιουργηθούν οι νομικές προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούμε και εντός των ε, ε, εδαφικών εδάτων της Λιβύης. Για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και θα χρειαστεί επίσης νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα πρέπει όμως επίσης να λυθούν και τα νομικά θέματα. Σήμερα όσοι διασώζονται παραδίδονται στην Ιταλία, στις Ιταλικές αρχές αλλά και φυσικά ισχύει αυστηρά η αρχή της μη επαναπροώθησης. Ε, αλλά ε, όταν θα πια εντός ε, των ε, υδάτων της Λιβύης δεν θα ισχύει πια αυτό. Εάν λοιπόν συλλάβουμε ε, μετανάστες θα, θα τους φέρουμε στην Ιταλία διότι ισχύει η αρχή της μη επαναπροώθησης αλλά τους διακινητές δεν θα μπορούμε να τους μεταφέρουμε στην Ιταλία. Και δεν μπορούμε να τους παραδώσουμε ούτε στη Λιβύη, διότι δεν υπάρχει σχετική συμφωνία ανάμεσα στη Λιβύη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να απελευθερώνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση προτού να έχει επιληθεί αυτό το νομικό πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι θα αργήσουμε να δούμε λύση στο θέμα αυτό στη Λιβύη. Οι ε, κρατούμενοι δεν ε, έχουν τις συνθήκες που θέλουμε να εφαρμόζονται. Η Ιταλία σήμερα ε, ε, προσπαθεί να ε, διώκονται οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες προέλευσής τους ή θα μπορούσε να ισχύσει το πρότυπο Αταλάντα ώστε να μεταφέρονται σε τρίτες χώρες. Ελπίζω το θέμα αυτό να επιληθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάντως αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εργαζόμαστε εκτός των υδάτων της Λιβύης. Και αυτά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, σήμερα. Έχουμε ένα σκάφος ε, ιταλικό, δύο γερμανικά, ε, μία ισπανική φρεγάτα και ένα πλοίο των του, του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε επίσης κάποια άλλα σκάφη και ένα υποβρύχιο. Για πρώτη φορά λοιπόν Έχουμε ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη στο κέντρο της Μεσογείου με αυξανόμενη παρουσία. Έχω κάνει πολλά ταξίδια, έχω συναντηθεί με πολλούς διεθνείς οργανισμούς σε διάφορες χώρες για να εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε για να εξηγήσω και τι δεν κάνουμε, τι δεν καλύπτεται από τις ε, δραστηριότητές μας. Η επιχείρησή μας ε, είναι πολύ γνωστή σήμερα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε δημιουργήσει ένα φόρουμ που λέγεται Segment, όπου συναντώνται όλες οι χώρες ε, και συζητούν τη δυνατότητα εξέβρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης. Η πρώτη συνάντηση έγινε τον Νοέμβριο, η επόμενη θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Οχτώ ομάδες εργασίας ε, εργάζονται με στόχο να προτείνουν λύσεις για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σήμερα, όπως σας είπα, ε, όσοι διασώζονται στη θάλασσα μεταφέρονται στην Ιταλία. Το Ιταλικό ε, Υπουργείο Εσωτερικών ε, καθορίζει τον ε, λιμένα όπου φέρνουμε τους ανθρώπους αυτούς και εφαρμόζουμε αυστηρά την αρχή της μη επαναπροώθησης. Έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, έχουμε συνδέσμους ε, της Frontex πάνω στα σκάφη που συμβολεύουν τους πλοιάρχους. Και είναι υψής της σημασίας η καλή συνεργασία. Συνεργαζόμαστε στενά, διότι θέλουμε να ανακόψουμε τις δραστηριότητες των διακινητών. Ουσιαστικά πρόκειται για αστυνομική επιχείρηση με στρατιωτικά μέσα. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τον Ιταλό ισαγγελέα για το οργανωμένο έγκλημα. Και με την Interpol προβλέπεται ανάλογη προσπάθεια. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ε, την UNHCR, την UNICEF και άλλους που ε, εκπαιδεύουν τα ε, πληρώματά μας και επίσης έχουμε κάποιες πρότυπες μεθόδους εργασίας και εγχειρίδια σχετικά με την μεταχείριση μεταναστών. Η συνεργασία αυτή είναι υψής της σημασίας. Η UNAFORMED έχει παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσματα και νομίζω ότι αποτελεί την απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει κάτι συγκεκριμένο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 24 κράτη-μέλη συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Έχουμε καλύτερη κατανόηση των ε, μεθόδων των διακινητών, ε, έχουμε σώσει 12.000 ε, ανθρώπους, έχουμε συλλάβει 68 διακινητές ε, και έχουμε καταστρέψει 104 σκάφη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πονάβαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο στη συνέχεια, μπορείτε να, δείξετε, να κάνετε ένα νεύμα προς τη γραμματεία να σας καταγράψει. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ήθελα απλώς να πω η Σοφία είναι ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε σε ένα από τα πλοία μας, σε μια γερμανική φρεγάτα. Το παρατσούκλι της ε, φρεγάτας ήταν Σοφία και γι' αυτό δόθηκε αυτό το όνομα στην ε, επιχείρηση και είπα ότι η εκπρόσωπος θεώρησε ότι το καλύτερο όνομα για αυτή την επιχείρηση είναι πράγματι η Σοφία. Αυτή είναι η Σοφία πριν από ένα μήνα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πραγματικά δείχνει το περιεχόμενο της δράσης μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μωράης. Από την ε, Frontex επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ο κύριος ε, παρετέρος στην MED και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα επιχειρησιακών δράσεων, εκπαίδευση πληρωμάτων κτλ. Θα ακούσουμε από την ε, κυρία Στραζιέρη για τον ρόλο της ε, Frontex, αλλά φυσικά και για τους, τον κύριο Στραζιέρη για τους οργανισμούς αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Η συνάντηση αυτή μας καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει πια το σύστημα των στεγανών πυλώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω συναδέλφου με του οποίου συνεργαζόμουν του τελευταίου 12 μήνε, τον Ερικό Καντίνο, με τον οποίο εργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε για πάνω από 10 μήνε ή κάτι τέτοιο, και με τον Όλτριτ Μαρτίνου και τη Europol έχουμε μακρά συνεργασία γιατί οι φορείς αυτοί στον τομέα των θεμάτων δικαιοσύνης και εσωτερικών είναι φυσικοί εταίροι. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα και μόνο παραδείγματα δράσης και συνεργασίας που ο στόχος τους πάντα είναι να εξασφαλίσουν τον έλεγχο και την εξασφάλιση των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα στη συνέχεια να κλείσω με κάποια σχόλια για το ρόλο της Frontex στο μέλλον, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε επίγνωση. Ξέρουμε ότι τώρα υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την μελλοντική εντολή της Frontex. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, το παράδειγμα συνεργασίας με την Uniformed ίσως το ξέρετε ήδη, τα μέλη του Κοινοβουλίου ξέρουν πολύ καλά τα θέματα της Frontex, ίσως κάποιοι από εσά όμως δεν τα έχετε υπόψη σας. Ο κύριος Ρόλος, η κύρια αποστολή της Frontex, είναι ότι είναι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανήκαμε λοιπόν στον πρώτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επί τη βάση του κώδικα του Σέγγελ και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Frontex συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής πολιτικής, επομένως εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλοι εταίροι μας, όπως οι αποστολές CSDP και ΕΠΑ, είναι σε ένα άλλο πυλώνα ευρωπαϊκών πολιτικών. Παρά το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικές εντολές, παρά το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικό τεχνικό εξοπλισμό, μπορούμε να έχουμε ένα συμπληρωματικό ρόλο μεταξύ μας. Για παράδειγμα, με την UNAFOR, όπως ελέγχθη <clears throat> προηγουμένως, έχουμε συμφωνήσει να έχουμε αξιωματικούς συνδέσμους, να ανταλλάσσουμε αξιωματισμούς. <clears throat> Μπορούμε να έχουμε λοιπόν στην Κατάνια αξιωματικούς από την ε, UNAFOR που έρχονται στην Κατάνια, όπου και άλλοι φορείς όπως η UNAFOR έχουν εκπροσώπηση, επίσης Έχουμε αξιωματικούς συνδέσμους στην ναυαρχίδα της επιχείρησης Uniformed και επίσης έχουμε και ένα σύνδεσμο στο, στο αρχηγείο της Uniformed στην ε, Ρώμη. Ο στόχος αυτής της, αυτής της ανταλλαγής αξιωματικών συνδέσμου είναι να έχουμε σε πραγματικό χρόνο όσο καλύτερη ε, αλληλοπληροφόρηση και μια ενιαία εικόνα της κατάστασης. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητα λοιπόν αυτά και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και είναι απαραίτητα ιδίω σε επιχειρήσεις έρευνα και διάσωσης να ξέρουμε πού ακριβώς είναι τα πλοία μας και ποιος μπορεί το ταχύτερο δυνατό και πιο αποτελεσματικά να παρέμβει για τη διάσωση ζώων. Να υπογραμμίσω επίσης το γεγονός ότι υπάρχει και ανταλλαγή απόψεων στον τομέα της ανάλυσης κινδύνων. Αυτό είναι ένα σημαντικό τομέα δραστηριοτήτων. Στον πυρήνα της εντολή της η Frontex περιλαμβάνει και την εποπτεία των συνόρων και η Frontex στην Ιταλία έχει 10 πλοία περιπολίας. Έχουμε επίσης και πολιτικά αεροσκάφη που ασκούν αυτό το έργο όταν <clears throat> διακριβώνουμε την παρουσία ανθρώπων στη θάλασσα, τους ε, διασώσουμε ή εμείς οι UNAMFORMED και όταν τους αποβιβάσουμε τους πιέλουμε στα διάφορα hot spots, τους ε, ε, κάνουμε συνεντεύξεις μαζί τους, συλλέγουμε πληροφορίες και μαζεύουμε δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται στην Europol, Europol στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Επομένως, η Frontex είναι μια γέφυρα μεταξύ από τη μία πλευρά της EU ε, NAVFORMED που είναι μια στρατηγική επιχείρηση και από την πλευρά των εθνικών ε, διοκτικών και αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων αυτών στα εθνικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όταν πρόκειται για τη συνεργασία με την Europol, είναι σημαντική αυτή η συνεργασία γιατί όπως σας είπα είμαστε και οι δύο φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εσωτερικών και δικαστικών θεμάτων. Έχουμε κάποιες <clears throat> συμφωνίες συνεργασίας. Μαζί με τον ομόλογό μου το Δεκέμβριο υπέγραψα μια νέα συμφωνία για την συνεργασία μας που εστιάζει περισσότερο στην ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Έχουμε εκκινήσει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της δράσης της Frontex με όνομα Triana Trident και η λογική και η, ο στόχος αυτού του συστήματος, αυτής της συνεργασίας είναι να υπάρξει ένα είδος φιλτραρίσματος των εξωτερικών ε, συνόρων στα, σύνορα της Ευρωπα... στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όρια της ε, περιοχής ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό για να εξασφαλίσουμε την εντόπιση κινδύνων <clears throat> και φυσικά αυτό αφορά και το, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο και ενδεχομένω και τη τρομοκρατία. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εσωτερικά σύνορα όμω ω ένα φίλτρο γιατί δεν θέλουμε ορισμένα άτομα να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και το πρόβλημα των ξένων μαχητών οι οποίοι φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με την Ευρωπόλεμη, ε, αναπτύσσουμε μια διαδικασία συλλογής προσωπικών στοιχείων που εστιάζονται περισσότερο στην ε, εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων. <clears throat> δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανακρίνουμε κανένα γιατί δεν έχουμε δικαστικές εξουσίες, αλλά η Frontex έχει σαν στόχο και αποστολή να συλλέγει και να επιμερίζεται πληροφορίες με την EU Now δεν πρόκειται για προσωπικά στοιχεία. Έχουμε συμφωνήσει για κάποιες κοινέ διαδικασίες με την EU format για το πού θα υπάρχουν τα διάφορα πλοία μας. Έχουμε αποφασίσει να έχουμε ανταλλαγή στοιχείων για αξιολόγηση κινδύνου, αλλά δεν έχουμε καθόλου ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Αυτό γίνεται με τα κράτη-μέλη υποδοχής που στην περίπτωση αυτή είναι η Ιταλία. Αυτή λοιπόν είναι η γενική εικόνα της συνεργασίας μας. Αν μπορώ τώρα να περάσω σε κάποια καταληκτικά σχόλια. Όπως σας είπα, δεν έχουμε πια καθόλου χωριστούς πυλώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί όταν πρόκειται για την ε, εποπτεία των συνόρων ή την διαχείριση πρώτης έλευσης στα σύνορα, η κατάσταση στην ε, Λιβύη είναι τέτοια, ώστε με μη στρατιωτικά μέσα δεν θα μπορούσαμε να εποπτεύουμε την κατάσταση αυτή και αυτό ισχύει, θα μπορούσε να ισχύει στο μέλλον και σε άλλες περιοχές όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε με κράτη τα οποία έχουν δυσλειτουργίες, κάτι που έχουν αστοχήσει. Στη Λιβύη βέβαια, όπως ξέρετε δεν έχουμε τέρους, αυτό μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον, αλλά η κατάσταση ασφαλείας για το προσωπικό μας δεν επιτρέπει να έχουμε στρα... να μη στρατιωτικό προσωπικό και μέσα στη Λιβύη. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες περιπτώσεις όταν η, τα πλοία ή ο εξοπλισμός της Frontex χρησιμοποιείται για έλεγχο στις ακτές της Λιβύης, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε επιθέσεις, πυροβολισμούς κτλ. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να μας προστατεύσουν στρατιωτικές δυνάμεις. Συγχρόνως όμως, Υπάρχουν και κάποιες αποστολές που είναι καθαρά εφαρμογής του νόμου για στόχους εσωτερικής ασφάλειας και έχω στο μυαλό μου εδώ την Europol και η Frontex βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί θα πρέπει να παίξει τον απαραίτητο ρόλο για να δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται και η Europol. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το μελλοντικό σκοπό και την εντολή <clears throat> της ε, Frontex, η πρόταση της Κομισιόν είναι να διευρύνει την εντολή μας και στον τομέα της ακτοφυλακής, αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία με τις ε, αρχές εφαρμογής του νόμου και αυτό το οποίο θέλουμε τώρα να δημιουργήσουμε επιτόπου στην Ιταλία ένα πολύ καλό παράδειγμα. Να σας αναφέρω επίσης και σε σχέση με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, να αναφέρω ότι αυτά που κάνουμε μαζί με τη Europol στα ελληνικά hotspots, ιδίως, εκεί σε αυτήν την πρώτη γραμμή η Frontex έχει αξιωματικούς οι οποίοι υποστηρίζουν την Ελλάδα για τον έλεγχο ασφαλείας επί τη βάση του συστήματος πληροφόρησης του Σέγγεν και σε ένα δεύτερο επίπεδο η Europol μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία περιπτώσεων που είναι ύποπτες αν αναδυθούν τέτοιες περιπτώσεις. αν επέχουν κίνδυνο τα άτομα, αν επέχουν κάποια απειλή. Αυτά κάνουμε λοιπόν σε καθημερινή βάση, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό μέλλον για τη Frontex και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όλα αυτά αφορούν μη στρατιωτικέ αποστολέ. Θα ήθελα λοιπόν να πω αυτά τα οποία λέχθηκαν και προηγουμένω. Πρόκειται για μια πολιτική και όχι στρατιωτική επιχείρηση, η διαχείριση των συνόρων και υπάρχει μια ε, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Frontex για τον σκοπό αυτό, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να συνεργαστούμε και με άλλες υπηρεσίες και φορείς, παραδείγματος με ευρωπαϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις και επειδή υπάρχει εδώ και ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, <clears throat> θέλω να πω ότι η Frontex μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχει αναπτύξει και συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Λετζέρη. Αναφερθήκατε πολλές φορές στην Ευρωπόλ και στη συνεργασία και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της ε, λαθρείας διακίνησης δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο οπότε θέλουμε να μάθουμε περισσότερα τι γίνεται, ε, τι γίνεται με τις εργασίες στο νέο κέντρο σε σχέση με την Ευρωπόλ. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Κύρια Πρόεδρε, αξιότιμοι καλεσμένοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπόλ ε, αισθάνεται πολύ ικανοποιημένη που την καλέστε εδώ για να συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση, ώστε να σας ε, δώσει τις τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με τον ρόλο που εμείς ε, ε, παίζουμε στην αντιμετώπιση των λαθρέων διακινητών. Η ζωή μου είναι λίγο ευκολότερη. Η ζωή μου εμένα είναι λίγο ευκολότερη ακούγοντας τον κύριο Λετζέρη καταλαβαίνει κανείς πόσο στενά συνεργάζονται αυτοί οι δύο οργανισμοί. Και θα αναφερθώ και εγώ στη συνεργασία αυτή, αλλά θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για τις τάσεις που παρατηρούνται ε, βάσει των κοινών μας ε, αξιολογήσεων με την Interpol. Έτσι δημιουργήσαμε το κέντρο κατά της λαθρές διακίνησης ε, μεταναστών τον Ιανουάριο φέτος και μετά θα σας παρουσιάσω τις ε, δυνατότητες, τους μηχανισμούς που έχουμε, που προσφέρουμε ε, και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα κράτη-μέλη. Αλλά να μην ξεχάσω πρώτον τους χαιρετισμούς του κ. Wainwright, ο οποίος την τελευταία στιγμή χρειάστηκε να πάει στο Λονδίνο διότι εκεί υπάρχει μια διάσκεψη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οπότε σας στέλνει χαιρετισμού. Εγώ τον αντικαθιστώ, είμαι αναπληρωτής διευθυντής ε, εδώ και για 27 χρόνια υπήρξα αστυνομικό και υπήρξα και αρχηγός της αστυνομίας στη Τσεχική Δημοκρατία πριν να ε, μετατεθώ στην Ευρωπόλ. Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή βρισκόμαστε έντο του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την υποστήριξή σας κατά τη δημιουργία του Κέντρου Αντιμετώπισης Λαθρείας Διακίνησης Μεταναστών. Μας υποστηρίξατε για να λάβουμε επαρκή χρηματοδότηση. Κάτι που μας βοήθησε πολύ στο να το κάνουμε πραγματικότητα. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε εδώ μαζί με άλλους συναδέλφους και εκπροσώπους σημαντικών οργανισμών που όλοι σε κάποιο βαθμό ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Η άποψή τους λοιπόν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και προσπαθώ να βρω και πώς συμπληρώνουμε ένα τον άλλον. Γιατί ναι, πρέπει να ακολουθούμε με ε, τις εντολές που έχουμε ο καθένας, αλλά πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε και σημεία επαφή, σύνδεσης και τρόπους συνεργασίας μεταξύ μας. Όσον αφορά τις τάσει της λαθρέα διακίνησης ε, μεταναστών, όπως ανέφερα στην κοινή μα συνεργασία με την Ευρωπόλα, αυτή η απροσδόκητη εισρωή μεταναστών άλλαξε το ποινικό τοπίο. Άλλαξε το τοπίο, το, την εικόνα των εγκληματιών ουσιαστικά. Πρόκειται για δίκτυα που ασχολούνταν σε άλλους τομεί και απλά επέκτηναν τι δραστηριότητε του, οι οποίε είναι επικερδεί και με χαμηλότερο κίνδυνο. Αυτέ οι δραστηριότητε λοιπόν ε, διακίνηση μεταναστών που να αναπτύξουν ένα νέο εγκληματικό μοντέλο. Μετά από 1.500 περίπου συνεντεύξεις μεταναστών, ε, ανακαλύψαμε ότι το 90% των μεταναστών που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν υπηρεσίες διευκόλυνσης στις περισσότερες περιπτώσεις από εγκληματικά δίκτυα. Ταυτόχρονα ε, έτσι ε, σχηματίζεται η εικόνα των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει, ε, έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Απόψη χρηματική εκτιμάται ότι τα εγκληματικά δίκτυα, αυτοί οι διακινητές, παρήγαγαν μεταξύ τριών και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 μόνο. Η δραστηριότητα αυτή λοιπόν υπήρξε πολύ ελκυστική το 2015 και βλέπουμε ότι συνεχίζεται το 2016 και αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Η αγορά αυτή θεωρείται μία από τις πλέον ταχαίως αναπτυσσόμενες εγκληματικές αγορές από ευρωπαϊκή άποψη το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο ονομάζεται έγκλημα ως υπηρεσία ε, περιλαμβάνει την εκδοση διαβατηρίων, ε, την παροχή μέσων μεταφοράς, ε, σκαφών, ε, μετάβαση χρημάτων, διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από ειδικευμένες ομάδες εγκληματιών. Επίσης έχουν δημιουργήσει και μια νομική δομή, δομή νομικών υπηρεσιών που παρέχονται ε, σε περιπτώσεις φυλάκισης ή και για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούνται επίσης ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Προσελκύουν ανθρώπους ε, τους οποίους προσλαμβάνουν μέσω των ε, μέσω κοινωνικών δικτύων, δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου κτλ. Οι δομέ αυτέ οι εγκληματικέ ασχολούνται και με την ε, επωνομαζόμενη δευτερεύουσα κατανομή των μεταναστών, διανομή των μεταναστών σε διάφορε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφοροι ε, παραγόντες σε διάφορε φάσει, ξεκινώντα από τους υπεύθυνου για τις προσλήψεις, ελαφρίους διακινητές, ε, άλλου που ασχολούνται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τη μεταφορά κονδυλίων. Και ταυτόχρονα κάτι σημαντικό που σχετίζεται με τους μετανάστες είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους πολύ ευάλωτους που αποτελούν το αντικείμενο εκμετάλλευση με διάφορους τρόπους, πορνεία, ε, διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Και αυτό σχετίζεται με άλλο ένα ενδιαφέρον έβριμο ότι αυτές οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ε, ασχολούνται με πολλές διαφορετικές μορφές εγκλημάτων και βλέπουμε τις συνδέσεις μεταξύ της διευκόλυνσης, της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της εμπορίας ναρκωτικών, αλλά βλέπουμε και συνδέσεις με την τρομοκρατία. Θα επανέλθω αργότερα σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις πιθανές ε, σχέσεις με την τρομοκρατία και ε, Θέλω να αναφέρω ένα κέντρο που δημιουργήθηκε πρόσφατα, το, κέντρο, το αντιτρομοκρατικό κέντρο, το οποίο συγχωνεύει ουσιαστικά κάποιες υπηρεσίες για να παρέχει υποστήριξη στα κράτη-μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση του τρομοκρατίας. Όταν εστιαζόμαστε σε αλλοδαπούς μαχητές, σε ανθρώπους που αποτελούν ε, ε, ισχυρή απειλή, εστιαζόμαστε σε οικονομικές πληροφορίες και σε άλλες πληροφορίες διότι ιστορικά δεν υπήρχαν ε, σχέσεις μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο σήμερα όμως αλλάζει. Το, οι, δραστηριότητες, οι σοβαρές δραστηριότητες σοβαρών εγκλημάτων χρησιμοποιούν ε, χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τις ε, πιθανές τρομοκρατικές δραστηριότητες. Γι' αυτό η σύνδεση αυτή είναι πολύ σημαντική και είναι πλέον ορατή η σύνδεση μεταξύ της παρανομής μετανάστευσης και της ε, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Η δημιουργία του κέντρου για τους μετανάστες το Φεβρουάριο, δεν τον γνωρίζουν, ε, αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία σε συνδυασμό με την επιχείρηση ΜΑΡΕ που στήθηκε το 2015 και εστιάστηκε στον εντοπισμό και την αποσάρθρωση ομάδων λαθρέας διακίνησης στη Μεσόγειο ε, βάσει αναλυτών και απεσπασμένων ε, εμπειρογνωμόνων από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο στη Μεσόγειο. Εμείς υποστηρίξαμε πολλές επιχειρήσεις. Έχω δύο σύντομα παραδείγματα. Η επιχείρηση Μαχμού που ολοκληρώθηκε πέρυσι το Δεκέμβριο που διεξήχθη σε διάφορες ε, χώρες ταυτόχρονα Αυστρία, Σουηδία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα 23 συλλήψεις διακινητών ε, Συρίων, Ελλήνων και Παλαιστίνιων πολιτών. Η επιχείρηση Τάνταλου τον Νοέμβριο πέρυσι όταν αλμανικές ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος διακινούσαν λαθρέα μετανάστες και αυτό κατέληξε στη σύλληψη 8 ατόμων ε, το οποίο επιτευχθεί χάρη σε πολλέ κατοικών έρευνε. Όσον αφορά τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, 40.000 περίπου υπόπτους για διακίνηση ε, παράτυπων μεταναστών, έχουμε αποθηκευμένους βάσεις δεδομένων μας, έχουμε περίπου, πληροφορίες για περίπου 100 ύποπτα σκάφη, έχουμε υποστηρίξει 1.500 επιχειρήσεις κατά το 2015 και όπως ανέφερε ο κύριος Λετζέρη συμβάλαμε στην περιφερειακή task force ε, στην Ιταλία και στην Ελλάδα όπου έχουμε στείλει συναδέλφους και αυτό το κέντρο αντιμετώπισης Λαθρίας διακίνησης μεταναστών αποτελεί πλέον ένα σημείο επαφής, μια πλατφόρμα και για άλλους εταίρους τους οποίους θεωρούμε σημαντικούς ε, για τη συνεργασία μας, Interpol, Frontex, UNFOS, ακόμη και το ΝΑΤΟ. Το Magnet Smuggling Center, το κέντρο αυτό, έχει δημιουργήσει περαιτέρω θέσεις, έχουμε ενισχύσει τις ε, δυνατότητες ανάλυσης, έχουμε περισσότερες, ε, περισσότερες δυνατότητες ανάλυσης των ε, εγκληματικών πληροφοριών, πληροφορίες που λαμβάνουμε και από διάφορα μέρη όπου βρίσκεται η Frontex όταν δηλαδή συλλαμβάνεται κάποιον, μαθαίνουμε κατά πόσο σχετίζεται με τρομοκρατία ή σοβαρό έγκλημα. Έτσι, οι πληροφορίες ε, ε, αυτές είναι πολύ σημαντικές ε, που έρχονται από τα σημεία που διεξάγονται οι επιχειρήσεις μας βοηθούν να αναλύσουμε την εικόνα και να κατανοήσουμε την εικόνα του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Στο κέντρο ε, στο τρομοκρατικό κέντρο έχουμε και μια μονάδα που επισημαίνει και εντοπίζει τους ε, ε, τρομοκράτες και τρομοκρατικό περιεχόμενο επίσης είτε στα μέσα κοινωνικά εις δικτύωσης είτε σε ιστοσελίδες. Το ίδιο μπορεί να κάνει και για τη διακίνηση, τη λαθρεία διακίνηση μεταναστών. Μπορεί να εντοπίσει σχετικές ιστοσελίδες ή λογαριασμού σε μέσα κοινωνική δικτύωση ε, που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση ε, της παράτυπη μετανάστευση. Τελευταίο, να διευκρινίσω, εγώ είμαι αστυνόμο και μερικές φορές ε, ε, χάνω την εικόνα των απτών αποτελεσμάτων. Γιατί εσείς, ξέρετε, βρίσκεστε στο μέτωπο. Εμείς Έχουμε ως κύριο στόχο να επεξεργαζόμαστε δεδομένα, να τα συμπληρώνουμε, να σας παρέχουμε υποστήριξη και αναλύσεις. Αλλά πρόσφατα δεν συντονίζουμε τις δραστηριότητε μας μόνο από τα κεντρικά. Ακολουθούμε και την απόφαση του Συμβουλίου για τους ε, προσκεκλημένους εξωματούχους και τώρα έχουμε αναπτύξει αυτή τη αυτό τον ορισμό και έχουμε αυτή την προτεραιότητα, τη νέα προτεραιότητα να έχουμε απεσπασμένους ε, ε, αξιωματικούς ε, που αμείβονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για, τις για τους δευτερεύοντες ελέγχους ασφαλείας. Δηλαδή έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και απλά επαληθεύουν την ορθότητα των δεδομένων. Τέλος, όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και τους διεθνείς οργανισμούς, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και ειδικότερα για όσους δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο. Εμείς στην Ευρωπόλ ενδιαφερόμαστε για όλα τα είδη πληροφοριών που σχετίζονται με τους διακινητές. Οτιδήποτε μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και τις αναλύσεις μας. Πληροφορίες που ούτως άλλως στέλνουμε ξανά στα κράτη-μέλη, τα οποία είναι αρμόδια να ε, βάλουν φυλακή αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Αυτά από πλευράς μου και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. final speaker. Και έχουμε τελευταία ομιλήτρια την ε, πρέσβυρα Φρανσέσκα Ταρτιόλη ε, από τον ΝΑΤΟ. Δέκα λεπτά παρακαλώ το πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει σε αυτήν την κοινή ακρόαση. Ακούσαμε ότι η η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ε, μεγαλύτερη ε, κρίση προσφύγων και μεταναστών ε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Ε, αποκτήσατε μια εικόνα του τι γίνεται από τους προηγούμενους ομιλητές. Ε, θα ήθελα ε, να ξεκαθαρίσω ότι το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται επικεφαλής των προσπαθειών αυτών, αλλά προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Frontex και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Η συμμετοχή του ΝΑΤΟ αποφασίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου από τους Υπουργούς Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και συμφώνησαν να ανταποκριθούν θετικά στις προτάσεις Γερμανίας, Ελλάδας και Τουρκίας ε, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ε, με συμμετοχή στην μεγάλη διεθνή προσπάθεια να ανακοπούν οι πορείες των διακινητών στην Μεσόγειο. Η το ΝΑΤΟ λοιπόν εποπτεύει στο Αιγαίο σε συνεργασία με ε, την Frontex μεταξύ άλλων. Κατέστασαν λοιπόν ε, τα σκάφη του ΝΑΤΟ δύο μέρες ε, μετά την λήψη της υπουργικής απόφασης και μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες τα σκάφη του ΝΑΤΟ περιπολούν σε συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου μεταξύ άλλων εδαφικά, στα εδαφικά ύδατα Ελλάδα και Τουρκίας. Ε, τα σκάφη μας έχουν συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και από τις ελληνικές ε, και ε, τουρκικές ε, αρχές, τις ακτοφυλακές, καθώς και από το ΝΑΤΟ. Οι εργασίες πραγματοποιούνται ομαλά, υπάρχουν ρυθμίσεις για συνδέσμους ΝΑΤΟ και Frontex, καθώς και σε συνεργασία με την ομάδα που δραστηριοποιείται στο Αιγαίο. Και ακριβώς ε, έτσι φαίνεται πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μπορούν να συνεργαστούν με αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη μας. Αυτές οι ρυθμίσεις σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο συμφωνήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τον ε, περιορισμένο και συγκεκριμένο ρόλο του ΝΑΤΟ. Η συμβολή του ΝΑΤΟ είναι σημαντική και μεγάλης ε, αξίας ε, δεδομένης δεδομένων των δυνατοτήτων του. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ συγκεκριμένη η προσπάθεια αυτή. Δεν υποκαθιστούμε τις εθνικές δυνατότητες, αλλά βοηθάμε τις εθνικές, ελληνικές και τουρκικές αρχές να εκτελέσουν τα καθήκοντά του με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, είδαμε σχεδόν ε, κάθε μέρα ε, περιπτώσεις εντοπισμού σκαφών με μετανάστες. Έχουμε διαβάσει τις πληροφορίες αυτές στις εθνικές αρχές της Ελλάδας, της Τουρκίας και στην Frontex και κατόπιν έχει αναλυφθεί η δράση από πλευράς αυτών για να ανακοπεί η πορεία των σκαφών αυτών. Έχουμε βοηθήσει στην βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ε, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που μπορεί να επηρεάσει τις ε, μεταναστευτικές και προσφυγικές ζωές, ώστε όσο η παρουσία του ΝΑΤΟ κατά τη γνώμη μου ήδη ε, ε, έχει παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα και έχει αποτρέψει το οργανωμένο έγκλημα ανάμεσα στις ακτές Τουρκίας και Ελλάδας. το ΝΑΤΟ θα εξετάσει πολύ σύντομα πώς θα μπορέσει να διατηρήσει τις δραστηριότητε αυτές ε, μακροπρόθεσμα. Ο ε, υπονάβαρχος ε, Τρεντετίνο αναφέρθηκε ε, στο θέμα αυτό πριν. Ε, τώρα λοιπόν η επιχείρησή μας αυτή γίνεται επιχείρηση ασφάλεια στη θάλασσα, κάτι δηλαδή ε, που θα μπορεί να καλύψει περισσότερα καθήκοντα από αυτά που εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Κάτι τέτοιο θα μπορεί να επιτευχθεί, αυτό είναι ο στόχος τουλάχιστον, μέχρι την επόμενη διασκέψη κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία τον Ιούλιο και η επιχείρηση Endeavor θα μπορέσει να αποτελέσει πλαίσιο και για τον μελλοντικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων ε, του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Εξετάζοντα ε, τι προκλήσει ε, που αντιμετωπίζονται στο Αιγαίο, θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο Ναύαρχο Κρεντεντίνο αυτά που έχουμε πετύχει με την επιχείρηση Σοφία ήταν πολύ σημαντικά και ελπίζω ότι θα μπορέσει να διευρυνθεί αυτή η συνεργασία και στο μέλλον. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε ε, τις γενικότερες διαστάσεις ε, των, ε, της προσφυγικής κρίσης σε άλλες περιοχές πέρα από το Αιγαίο. Φυσικά θα διατηρήσουμε και, στενές, ε, και τη στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κλείσω με μια παρατήρηση που έχει να κάνει με τις νομικές πτυχές, κάτι που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σας. Η καθοδήγηση προς τους πλοιάρχους στο Αιγαίο είναι ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ και η κινητοποίηση δυνάμεων του ΝΑΤΟ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο κατά περίπτωση. Κάθε κράτος που συμμετέχει δεσμεύεται να τηρεί το εθνικό και διεθνές δίκαιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, να σεβόμαστε την αρχή της μη επαναπροώθηση, της διάσωσης στη θάλασσα κλπ. Θα ήθελα να κλείσω εδώ. Επτά λεπτά μίλησα. Ε, βλέπετε, στρατιωτική πειθαρχία έχω και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ διπλωματικά το να χρησιμοποιήσετε λιγότερο χρόνο όταν όλοι αρχίζουμε να κουράζονται η ανθρώπινη κατάσταση αυτή δεν μπορεί κανείς να συλλέξει και να κατανοήσει τόση πολλή πληροφορία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση. καθώ μιλούσατε εγώ σκεφτόμουν ότι ακούγαμε την φωνή του ΝΑΤΟ. Ένα από του λόγου για τον οποίο η κυρία Φωτίγα πρότεινε να γίνει αυτή η κοινή ακρόαση είναι ότι γιατί μερικέ εβδομάδε υπήρχε πολλή ανησυχία για το γεγονό ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ φορέων υψηλού επίπεδου που οι επιτροπές μας είναι αρμόδιοι για την εποπτεία τους και έχει συνεχιστεί αυτή η συνεργασία τις τελευταίες εβδομάδες. Εμείς ως μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών θέλουμε να έχουμε λεπτομεριακές δομές λογοθεσίας από φορείς όπως η Europol, η Frontex, η Eurojust και νομίζω και η δική σας Επιτροπή, η Υποεπιτροπή έχει τέτοια, τέτοια ανάγκη. Όταν υπάρχει λοιπόν ενισχυμένη συνεργασία και δεν είναι φανερό ποιε είναι οι δομέ λογοδοσία, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σωστό <clears throat> να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει πραγματικά μεγάλη εστίαση στο θέμα του πώ λειτουργεί η λογοδοσία για την επιχείρηση αυτή στη Μεσόγειο. Πολύ χάρηκα λοιπόν που άκουσα τους ομιλητές μας ο Κρίσον Έλερν, αυτός ο οποίος ζήτησε πρώτο το λόγο. Παρακαλώ συνάδελφοι να παραμείνετε στα δύο-τρία λεπτά το πολύ. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σταματήσω πάντα. Κρίσεν, είσαι εσύ ο πρώτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Να ευχαριστήσω και τους δύο συμπρόεδρους και τις γραμματείες που οργάνωσαν αυτήν την ακρόαση. Νομίζω ότι ήταν καιρό να γίνει κάτι τέτοιο και υπήρξε μια συναντήληψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο όχι μέσα από στεγανά, αλλά να συνδυάσουμε και την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση του προβλήματος αυτού. Εγώ έχω δημοσιεύσει ένα βιβλίο για την μακρά πορεία προς την Ευρώπη και στην διάρκεια της έρευνάς μου για αυτό το βιβλίο ήταν φανερό ότι έχουμε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι Ε, έχουν και κάποια σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε αυτούς τους τρεις πυλώνες, αν θέλετε. Αλλά ας μπούμε στις λεπτομέρειες λίγο περισσότερο. Αναφέρατε την ανάγκη για συνεργασία σε υψηλό επίπεδο. Αναφερθήκατε στις συμφωνίες οι οποίες έχουν συναυθεί. Πώς γίνεται όμως στην πράξη. Έχω μία συγκεκριμένη μελέτη που αφορά ένα κοινό πρόγραμμα μετάφρασης. Παίρνουμε στοιχεία από την Βόρεια Αφρική στα αραβικά, το οποίο μεταφράζεται πρώτα στη Γαλλία προς τα γαλλικά και μετά από τη Γαλλία περνάει στα αγγλικά και τα γερμανικά και μετά διανέμεται στα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν 16 υπηρεσίες πληροφορικής και μετάφρασης πολλές φορές ένα όνομα το οποίο έχει μεταφερθεί από τα αραβικά ή τουλάχιστον μια λέξη της αργό στα αραβικά έχει 12 ή παραπάνω διαφορετικές εκδοχές. Αυτό μου είπαν τουλάχιστον οι υπηρεσίες μετάφρασης. Και εδώ τίθεται το θέμα της ανταλλαγής δεδομένων. Τα συστήματα ταυτοποίησης, οι εικόνες από τους δορυφόρους. Η πραγματική λοιπόν πρόκληση είναι η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων αυτών των υπηρεσιών. Και από την οπτική γωνία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η ανάγκη το Κοινοβούλιο να έχει μια σφαιρική εικόνα, μια συνολική εποπτεία ε, των ενεργειών αυτών των υπηρεσιών. Ποια είναι η δική μας εμπειρία στον τομέα αυτό και τι θεωρείτε ότι λείπει από τη συνεργασία αυτή. Μίλησα για το σύστημα μετάφραση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανάγκε τεχνικού χαρακτήρα. Μπορείτε να πείτε κάτι περισσότερο για τα θέματα αυτά και το δεύτερο μου ερώτημα. Μπορεί να σας φανεί λίγο παράξενο στο πρίσμα της ασφάλειας. Είναι το θέμα της επικοινωνίας. Ένα παράδειγμα είναι το ότι μετά από τη διασύψη κορυφής και τα τελικά λόγια που έκανε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής του Συμβουλίου πέρασαν αμέσως στην Ιγυρία, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία αντιδράσεις αντιδράσει σε αυτά τα λόγια από τα κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάποια εποπτεία των επικοινωνιών στα κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης ούτε σε σχέση με την τρομοκρατία αλλά ούτε και στο πλαίσιο της ε, οργάνωσης της λαθρεμπορίας ανθρώπων. <clears throat> Επί τη βάση των πληροφοριών που έχουμε πάρει από εσά, ένα τρίτο του ΑΕΠ της Λιβύης περίπου αφορά την διακίνηση ανθρώπων. Δεν μιλάω για τα χωριά, <clears throat> δεν αναφέρομαι σε μικρές εγκληματικές οργανώσεις. Ακόμα και η Ιταλική μαφία θα το ζήλευε αυτό το 1 τρίτο του συνολικού εισοδήματος μιας χώρας της Μεσογείου να προέρχεται από την λαθρεμπορία και τη διακίνηση ανθρώπων. Και εκεί η επικοινωνία, η διακίνηση πληροφοριών, η, η παραπληροφόρηση αν θέλετε, έχουν αυτήν την τεράστια αγορά. Γιατί οι πληροφορίε που βγαίνουν στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα διαδικτύωση μεταφράζονται σε παραγγελίε και προμήθειε για του διακινητέ. Πώ λοιπόν μπορούμε εμεί να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τη σωστή επικοινωνία, να αναφέρουμε τα θέματα που μα ενδιαφέρουν, να πληροφορήσουμε και να προειδοποιήσουμε. Ξέρουμε <clears throat> ότι, μα το έχουν πει οι ΜΚΟ, ότι οι εγκληματικέ οργανώσει δαπανούν σε μέσα επικοινωνίας 400 φορές περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε εμείς λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σωστή επικοινωνία, ίσως το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα τύχει λανθασμένης ερμηνείας, όπως γίνεται τώρα να ανοίξουν διακινητές σε ένα άλλο δρόμο, να αλλάζει η τιμή, από, η τιμή διακίνησης από την Αιγυπτό στην η Ιταλία μετά από τη διάσκεψη κορυφής ανέβηκε τρεις φορές. Αυτά είναι τα πρακτικά θέματα. Τι χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσετε να εμποδίσετε τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ. Η Άννα Γκάμις. Ναι. Καλώς ήλθατε. Και είναι πολύ θετικό να έχουμε τελικά αυτή την κοινή συνάντηση των Επιτροπών Σέντα και Λίμπε, ώστε να συγχωνεύσουμε ή καλύτερα να οδηγήσουμε σε σύγκληση τις δύο οπτικές γωνίες εσωτερικής και εξωτερικής πτυχής της ασφάλειας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστών τον ναύαρχο, τον υπονάβαρχο Κρεδεντίνο, αν θα μπορούσε να μας επιβεβαιώσει ότι το πλοίο αυτό το οποίο βούλιαξε με περίπου 100 άτομα από την Αιθιοπία και τη Σομαλία. 400 άτομα λέει η ομιλητή τώρα. Αν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι είναι κάτι τέτοιο, είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για ανθρώπους. Επίσης, ξέρω ότι έχετε τονίσει ότι αυτή η επιχείρηση της EU Nav4 η Σοφία είχε σαν πρώτο στόχο να εμποδίσει το έργο των διακινητών. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια, όπως είπατε και εσείς ήδη. Εγώ ήμουνα ε, μέλος μιας αποστολής που πήγε πρόσφατα στα αρχηγεία σας στην Ρώμη και ξέρω ότι υπάρχουν ε, κάποια όρια. Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε στα ύδατα της Λιβύης. Γι' αυτό οι διακινητές φέρνουν τα τους ε, πρόσφυγες στα όρια των χωρικών υδάτων της Λιβύης και μετά η Σοφία αναλαμβάνει να τους διασώσει. Είναι, όπως είπατε, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα το γεγονός ότι έχει σώσει πάνω από 12.000 ζωές σε ένα χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εντυπωσιακό και δημιουργείται μια πάρα πολύ σημαντική θετική φήμη. Αλλά τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα όταν έχει κλείσει ο δρόμος των Βαλκανίων γιατί όπως είπατε θα οδηγήσει μάλλον σε μια μετακίνηση των οδών των διακίνητων. Μας είπαν ότι υπάρχει ένας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος για να φτιάχνονται φουσκωτά στην Κίνα και τα οποία περνάνε μέσα από χώρες που υποτίθεται ότι είναι εταίροι περνάνε από την Τουρκία, φτάνουν στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και μεταφέρουν τους ε, ευάλωτους ανθρώπους προς την Ευρώπη μέσα από τη Μεσόγειο. Εγώ μόλις πήγα στην Κύπρο σε μια αποστολή πάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πήγα και στην Βόρεια Κύπρο ακόμα και είδα κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Ότι εκεί υπάρχει μια, ένας οικονομικός κλάδος ανθών εισαγωγής κοριτσιών από την Ιγυρία για πορνεία, προς όφελος των στρατιωτικών που βρίσκονται εκεί. Και αυτό γίνεται από τις στρατιωτικές αρχές στην Βόρεια Κύπρο. Η Europol κάνει μια προσπάθεια να ανοιχνεύσει πώς λειτουργούν αυτά τα δίκτυα, γιατί για πρώτη φορά έμαθα κάτι τέτοιο να συμβαίνει και μέσω σοκάρισε. Για τη Λιβύη είδα τη δήλωση της ε, εκπροσώπου της κυρίας Μογκερίνη μετά από τη συνάντησή της με τους Υπουργούς Άμυνας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να της δώσουμε υποστήριξη για οποιαδήποτε επιχείρηση φύλαξης των συνόρων, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και περισσότερο από μια απλή ενέργεια φύλαξης των συνόρων. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Συρία στο να υπάρξει μια ενιαία δίκηση για την φύλαξη των συνόρων. Γιατί χωρίς ενιαία δίκηση δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, δικαστικής εξουσίας και της απουσίας της υπάτης αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Και τέλος, να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε εν ώψη της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και ο κ. Βετζέρη επίσης θα μπορούσε να απαντήσει ποια είναι η άποψή σας ότι θα έπρεπε και τα και οι ναυτικέ δυνάμεις να... Είναι πολλά τα τέλο ε, που είπατε, λέει ο κύριο. Ε, μόλις ε, πήγα στην Λέσβο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι εκεί παρόν το ΝΑΤΟ, αν τηρεί τον εθνικό νόμο και γιατί δεν σταματάτε αυτές τις αποστολές ε, που αντίκυνται στο εθνικό δίκαιο της χώρας Ελλάδος και δεν υπάρχει καν συμφωνία για απελάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία. Οι, ε, οι απελάσεις της βίας είναι κατά του διεθνούς δικαίου. Δεν ε, με αγνοούν τόσο πολύ τα μέλη της ΛΥΜΠΕ, συνήθως. Λοιπόν, έχουμε περισσότερα μέλη της ΛΥΜΠΕ που ζήτησαν τον λόγο από τη μέλη της ΕΝΤΕ. Δεν ακούστηκε τι είπε η κυρία Γκόμες. Ευχαριστούμε, Άννα. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που λέτε. Ας πάρουμε ένα μέλος της ΕΔΗ, κύριε Βάτμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα φλαμανδικά, αν μου το επιτρέπετε. Στα Ολλανδικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπόλ ειδικότερα. Την επισκέφθηκα πριν από δύο εβδομάδες περίπου και συμμετείχα σε κάποιες ενδιαφέρουσες ακροάσεις και συζητήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Είχαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες διευκολύνονται λόγω αυτή του διαχωρισμού μεταξύ ε, εσωτερικής πολιτικής ασφαλείας και πολιτικής άμυνας και όλοι τονίζουν ότι είναι σημαντική ανταλλαγή δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την αντιμετώπιση της ε, προσφυγικής κρίσης. Και θέλω να ρωτήσω τι δυνατότητες έχετε εσείς όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι κρίσιμη σημασία για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Δεύτερον, η Frontex, η Europol και η Eurojust έχουν ε, δημιουργήσει τις Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Task Force στην Κατάνια και στον Πειραιά. Τι διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτές τις Task Force. Τι έχουν μάθει αυτοί, αυτοί οι τρεις οργανισμοί από αυτή τη συνεργασία. Και τρίτον, είχαμε κάποιες συνομιλίες με την Ευρωπόλ πριν από λίγες εβδομάδες και μου είπαν ότι τα τελωνία της Μάλτας κατάσχεσαν ένα σωρό φουσκότα που έρχονταν από την Κίνα και προορίζονταν για τη Λιβύη. για τους διακινητές ανθρώπων. Έτσι φέρνουν ανθρώπους στην Ευρώπη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αφήσαμε τα, ε, τα φουσκωτά αυτά να πάνε στη Λιβύα. Αλλά αυτό που σας ερωτώ είναι πώς μπορούμε να το σταματήσουμε όλο αυτό ώστε οι διακινητές ε, ανθρώπων να μην έχουν τα μέσα. Διότι το 90% των μεταναστών που έρχονται εδώ έρχονται ε, μέσω λαθρέας διακίνησης. Πρέπει λοιπόν να ε, δίνουμε την ε, καταπολέμηση αυτών των δικτύων. Κλείνω τώρα τον κατάλογο. Πολλοί κόσμοι ζητάει τον λόγο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Και παρακαλώ, περιοριστείτε σε δύο-τρία λεπτά. Ο κύριος Κέρκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα αντισταθώ στον πειρασμό να κάνω υπερβολικά πολλές ερωτήσεις που αφορούν τη, θέματα που αφορούν τη ΛΥΜΠΕ. Θα κάνω λοιπόν μια ερώτηση που δεν αφορά μόνο τη δική ενημέρωση, αλλά έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ. Θα με ενδιαφέρει να μάθω ε, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των ναυτικών μονάδων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ποια είναι η ε, δομή της διοίκησης. Η Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ έχει συναντηθεί για να συζητήσει όλα αυτά. Ε, πρόκειται για μια επιτροπή που φαίνεται να έπεσε σε χρηστία για πολύ καιρό, όπω έχω καταλάβει, και να μην λειτουργεί τόσο καλά όσο λειτουργούσε παλιότερα, ενώ αποτελούσε ένα στο κομμάτι των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Σε ποιο βαθμό λοιπόν είναι πλάκη αυτή η πολιτική επιτροπή σε αυτέ τι συζητήσει και ειδικότερα στην, στον καταμερισμό εξουσιών. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Και το δεύτερο, όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων. Εγώ πρόσφατα είχα την εμπειρία του PNR και τώρα του ACRES. Οι βάσεις δεδομένων της Eurodact, του ACRES και του συστημάτων SIS. Όλα αυτά στο πλαίσιο των προτάσεων για τα έξυπνα σύνορα. Να ρωτήσω σε ποιο βαθμό έχουμε φτάσει, αν μη τι άλλο, σε μια πολιτική συμφωνία, για να μην πω πρακτική συμφωνία για το πώ θα λειτουργήσει η διαλειτουργικότητα απόψη τεχνολογικών λειτουργιών αφενό, αφετέρου και όσον αφορά τη δομή διοίκηση και ελέγχου αυτών των δεδομένων. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σκόγια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την τόσο σημαντική και τόσο επίκαιρη κοινή ακρόαση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους μας για τα σχόλιά τους. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όταν είναι τόσο πολύπλοκη η πραγματικότητα, τόσο σε ό,τι αφορά τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κρατη αλλά και τους άλλους εμπλεκόμενους διεθνού διεθνείς εταίρους, χρειάζεται συνεργασία. Και συμφωνούμε και εμείς ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να είναι πιο έντονη δυνατή όχι μόνο γιατί αυτό απαιτεί η αποτελεσματικότητα, αλλά για να αποφύγουμε την αλληλοεπικάλυψη των ενεργειών. Τρία σημεία. Ο κύριος Κρεντεσιάνο, ο υπονόμος Κρεντεσιάνο, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Frontex και αναφέρθηκε στους ε, αξιωματικούς συνδέσμους και την ανάλυση των κινδύνων. Το ερώτημα μου είναι, αυτή η συνεργασία αφορά τις επιχειρήσεις της κοινέ επιχειρήσεις όπως η Σοφία. Αφορά λοιπόν η συνεργασία μόνο στους αξιωματικούς συνδέσμου και την ανάλυση κινδύνου ή αφορά και το συγκεκριμένο περιεχόμενο των ενεργειών. Δεύτερο ερώτημα. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Frontex και ιδιαίτερα στον αγώνα κατά των κατά της ε, λαθρεμπορίας ανθρωπίνων όντων. Αν λοιπόν θα μπορούσε να ευνοηθεί περισσότερο αυτή η κοινή ενέργεια με καλύτερη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών ή αν αυτό θα έπρεπε να είναι από την πλευρά της Frontex ή αν αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μια προτεραιότητα. Και για τον κύριο Ρετζέρη, θα ήθελα να ξέρω αυτή τη στιγμή για την Frontex ποιες είναι οι πιο μεγάλες αδυναμίες της Frontex στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι γίνεται όταν αλλάξουν οι ε, δρόμοι διακίνησης προς την κεντρική Μεσόγειο και τι θα γίνει όταν έχουμε τις τραγωδίες αυτές όπως αυτές που είδαμε με πάνω από 500 νεκρούς την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Carlos. Ευχαριστώ, Κάρλος. Ο κύριος Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι παρουσιάσεις και νομίζω ότι αποτελούν καλό παράδειγμα συνεργασίας και συμπληρωματικότητας ανάμεσα ε, στους διάφορους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς συνδέεται αυτή η τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή με το οργανωμένο έγκλημα. Είπατε ότι το 90% όσων ε, καταφάνουν στην Ευρώπη πλήρωσαν ε, και η Europol έχει περίπου 40.000 υπόπτους ε, λαθρεμπορίας ανθρώπων. Τι μας εμποδίζει να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους πρώτων ευθυνών τους είναι πρόβλημα ανταλλαγή δεδομένων, είναι πρόβλημα αξιόπιστων πληροφοριών για να ξεκινήσει η δίωξή του. Και επίσης, γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν καταφτάσει, οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον είχαν κάποια χρήματα. Τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν καθόλου χρήματα. Βρίσκονται ακόμα στις χώρες ε, προέλευσης και ε, απλά δεν βλέπουμε τι τραγωδία περνούν. Και έχω μια ερώτηση ε, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ διαφόρων εγκληματικών ομάδων στη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι ε, που καταφάνουν στην Ευρώπη έχουν ήδη ε, τηλέφωνα, αριθμούς τηλεφώνων ε, εγκληματικών ομάδων, διακινητών κλπ. Μας είπατε ότι έχετε εντοπίσει περίπου 230 σημεία στην Ευρώπη, κάποια από αυτά στη Στοκχόλμη. Και επίσης, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους διακινητές και τις τρομοκρατικές ομάδες πώς, τι ποσοστό των 6 δισεκατομμυρίων αυτών ε, χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. Επίσης, οι εξτρεμιστικές ομάδες ε, στην Αίγυπτο ε, βρίσκονται σε ε, έχουν κάποια σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Ο πρόεδρος, ναι, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό και η ISIS. Η κυρία Ιώταλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε για αυτή την ιδέα που είχατε να συζητήσουμε από κοινού οι δύο επιτροπές τα πολύ σημαντικά ζητήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό το λόγο θα κάνω μία ερώτηση μόνο. Μετά από το κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού και μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διάσωσης στην ε, Μεσόγειο έχετε πραγματοποιήσει αναλύσεις ε, για το κατά πόσο υπάρχουν νέες απειλές, ε, κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να βρεθούν νέες οδοί μέσω της Αλβανίας ή των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων και αν ναι, ποια είναι τα μέτρα και η πολιτική της Frontex και των υπολείπων ευρωπαϊκών οργανισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σκακέλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας αυτές. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, καταρχάς, όσον αφορά την ε, επιχείρηση UNAFOR. Από τη δική μας πλευρά, από πολιτικής πλευράς, είναι κάπως περίεργο το ότι στέλνουμε το στρατό ε, στους πρόσφυγες και μετανάστες. Ε, έχουμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ε, που ε, πρέπει να ανακόψει την ε, πορεία των διακινητών και έχουμε και την ε, UNAFOR που έχει να κάνει με την προστασία των συνόρων. Είναι περίεργο λοιπόν που στέλνουμε τώρα το στρατό ε, για πρόβλημα προσφυγικό. Αλλά ίσως και αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Όσον αφορά την UNAFOR, η προστασία των συνόρων δεν καλύπτεται από την ΚΕΠΑ. Και το άρθρο 43 της ε, Συνθήκη της Λισαβόνα, ε, λέει ότι μπορούμε να έχουμε ανθρωπιστικές αποστολές, όχι όμως ε, προστασία των συνόρων. Αυτό πολιτική πλευρά, από νομική πλευρά είναι κάπω αμφισβητήσιμη ή αλλω είναι καθήκον τη Frontex. Φαίνεται να υπάρχει τεράστια σύγχυση και από πολιτικής πλευράς, από νομικής πλευράς είναι κάπως αμφισβητήσιμη η κατάσταση. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό και κάποιες ερωτήσεις επίσης, κύριε υπονάβαρχε. Όταν ξεκινήσει η τρίτη φάση, θα φέρνετε τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες στην Ιταλία, ε, θα απελευθερώνετε τους ε, διακινητές επειδή δεν μπορούτε να, τους, να ασκήσετε δίωξη. Πού όμως, στην ανοιχτή θάλασσα, στη Λιβύη, και κυρίως πώς θα κάνετε τη διάκριση. Σώζετε κάποιους που κινδυνεύουν στη θάλασσα, θα τους πάτε στην Ιταλία, αλλά θα πείτε ότι α, αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι διακινητής, δεν υπάρχει όμως ε, δικαστική απόφαση. Πώς μπορείτε να το καθορίσετε αυτό, μπορεί να έχετε κάποια υποψία και μπορεί να έχετε και δίκιο, αλλά πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι πρόκειται για διακινητή διότι αυτό το άτομο δεν θα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τη θέση του, να αποδείξει ότι δεν είναι. Και πέρα από αυτό, εάν απελευθερώσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τότε πώς καταπολεμούμε την ε, ελαφριά διακίνηση αν τους απελευθερώνουμε πάλι. Και ερώτηση προς τον Άτο, όσον αφορά την επιχείρηση στο Αιγαίο. Λέτε ότι ενεργείται εντός ε, του ε, διεθνούς και εθνικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά εάν έχουμε σκάφος του το μη τουρκικό που βρίσκεται σε τουρκικά ύδατα και συλλέξει ε, πρόσφυγες, ε, πού θα τους μεταφέρει. Και τελευταία ερώτηση, διασυνοριακό έγκλημα και εσωτερική ασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει συζητηθεί πολύ, αλλά εμένα με μπερδεύει η Europol και η Frontex. Πού, πώς ε, γίνεται η διάκριση των εντολών σας και ιδιαίτερα όσον αφορά τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η Frontex πρέπει να διασφαλίσει την εσωτερική ασφάλεια. Έχουμε όμως ε, και την Europol, έχουμε το διασυνοριακό έγκλημα που αφορά και τους δύο οργανισμούς. Πώς γίνεται η διάκριση. Ελπίζω να μπορέσει το πάνελ να έχει το χρόνο να απαντήσει γιατί είχε αυτά τα θέματα της ε, νομικής βάσης και νομικής εντολής είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και η Άννα μου είπε ότι στο επόμενο πάνελ ορισμένα από αυτά τα νομικά θέματα θα αντιμετωπιστούν. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα με τις ακροάσεις, ότι πολλοί φεύγουν επειδή είναι πολύ απασχολημένοι. Είναι σημαντικό όμως να διευκρινιστεί ποιος κάνει τι και επί τη βάση ποιας εντολής. Η κυρία Βίνμπεργκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν εδώ σήμερα για να μας ενημερώσουν. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Ο Ντόναλτ είπε τις προάλλες ότι ε, είναι τρομακτικός ο αριθμός ε, των ε, ανθρώπων που έρχονται από την Λιβύη. Αλλά τι περιμέναμε άλλωστε. Εφόσον έκλεισε η οδός μέσω Τουρκίας, αναμενόμενο ήταν να αλλάξουν δρόμο. Όσον αφορά την Λιβύη, και τον περιορισμένο αριθμό σκαφών ε, των διακινητών. Ακούσαμε περίπου πριν ένα χρόνο ε, ότι κατάφεραν να ανακτήσουν τα σκάφη αυτά με όπλα κιόλα. Ε. Και τώρα μιλάμε για στρατιωτική παρέμβαση από το φθινόπωρο και μετά. Αλλά εδώ διαβάζω ότι ε, έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις ε, που μπορούν ε, να να εξετάσουν ποιοι βρίσκονται πάνω σε ένα πλοίο. Αλλά η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Πώς βλέπετε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τέλος, διότι έπρεπε να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών, ο κύριος Τσίδεο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω όλους για τις τόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Μερικά σύντομα ερωτήματα μέσα στα πλαίσια των τριών λεπτών ελπίζω. Πρώτο ερώτημα. Αν αφήσουμε ελεύθερους τους διακίνητες, Μήπως έχετε σκεφτεί να στρεφείτε, στραφείτε σε ορισμένα κράτη-μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη για να βρεθούν νομικά εργαλεία που θα εξασφαλίσουν ότι θα μείνουν στη φυλακή. Είναι σαφές που θα πάνε, ξέρουν που θα πάνε. Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι είναι οι οργανωτές των ταξιδιών αυτών και οργανώνουν, οργανώνουν την παράνομη <clears throat> είσοδο σε ξένο έδαφος. Υπάρχει λοιπόν νομική ευθύνη αυτών των ατόμων και αυτοί θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το γεγονός ότι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρωπίνων όντων. Δεύτερο ερώτημα. <coughs> Έρχομαι, στρέφομαι προς τον υπονάβαρχο Κρεντεντίνο. Ποιοι είναι οι νέοι εναλλακτικοί δρόμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διακίνητες. Με ενδιαφέρει το θέμα της μαύρης θάλασσας. Θεωρείτε ότι είναι ασφαλής η μαύρη θάλασσα ή είναι και αυτός ένας δυνητικός δρόμος για την ε, διακίνηση παράνομων μεταναστών. Επίσης θέλω να ξέρω ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τον αριθμό των πλοίων, το ποσοστό των πλοίων που ανακόπτεται. Και ένα τελευταίο σχόλιο και εδώ θα ήθελα να έχω κάποια σχόλια και από τον κύριο Μαρτίνου. Λέμε πολλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία νομίμων δρόμων μετανάστευσης ως ε, εναλλακτική λύση έναντι της τωρινής διακίνησης ανθρώπων. Αλλά ανοίξουν νόμιμοι δρόμοι, αυτοί που είναι οι σημερινοί διακινητές, θα έρθουν αύριο στην Ευρώπη για να οργανώσουν από εκεί, στην Ευρώπη, την παράνομη μαύρη εργασία. Ξέρουμε ότι η, η μαζική ανεργία συνοδεύεται από εγκληματικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται αυτούς που είναι έξω από το εργασιακό πλαίσιο. Αυτό έγινε στι ΗΠΑ όταν πήγε το μεταναστευτικό ρεύμα και συνδυασόταν με διαφθορά. Το ίδιο πράγμα κινδυνεύει να γίνει στην Ευρώπη ή όχι. Θα ήθελα να έχω τη δική σα άποψη αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να υπάρχει εκμετάλλευση αυτών των νεόφερτων στην Ευρώπη οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα φάση εγκληματικής δραστηριότητας. Πάω κατευθείαν στον κύριο Κρεντεντίνο, συγγνώμη που έχουμε ε, προχωρήσει τόσο πολύ στον χρόνο. Τρία-τέσσερα λεπτά μπορείτε να εστιαστείτε στα βασικά θέματα. Ε, αυτά που θα σας πω είναι μη επιβεβαιωμένα ε, ε, για το ατύχημα που είπατε, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Η Uniformed δεν αφορά τι επιχειρήσεις προστασίας, είναι μια στρατιωτική επιχείρηση και έχουμε σαφή εντολή καταπολέμησης των διακινητών στο κεντρική και ε, Μεσόγειο ώστε να αναχαιτήσουμε τα μοντέλα διακίνησης. Δεν έχει να κάνει με σύνοριοφυλακή. Όταν συλλαμβάνουμε διακινητέ εντό των λιβικών χωρικών υδάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να του απελευθερώσουμε στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να του φέρουμε στη Λιβύη και δεν μπορούμε να του δώσουμε, να τους παραδώσουμε στη Λιβύη, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Λιβύη. Απλά του απελευθερώνουμε. Αλλά αν χρειαστεί να κάνουμε μια επιχείρηση διάσωση, τότε όσοι συλλαμβάνουμε είναι μετανάστες δεν κάνουμε, θεωρούνται μετανάστες, δεν κάνουμε τις ερευνές ε, επί του σκάφους. Τους δίνουμε στις Ιταλικές αρχές όπου μαζί με τη Frontex βλέπουν ποιοι είναι διακινητές και ποιοι είναι μετανάστες και τι είδους μετανάστες. Φυσικά δεν προτείνω τη μετάβαση στη φάση 2 μέχρι ε, όσο του ελοκληρωθεί το νομικό ζήτημα. Θα παραμείνουμε στην πρώτη λοιπόν φάση μέχρι τότε. Για τις νέες πιθανές οδούς Νομίζω ότι με το κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού οι άνθρωποι θα αρχίσουν να έρχονται μέσω θαλάσσης από το Λίβανο, τη Σύρια, την Αίγυπτο, την Αίγυπτο και ίσως την Τουρκία. Και η Μαύρη Θάλασσα δεν καλύπτει τη δική μου επιχείρηση, οπότε δεν έχω πληροφορίε. Ασχολούμαι απλά με του μετανάστε που έρχονται από, την, από τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, τη Μεσόγειο. Η σχέση μας με τον ΝΑΤΟ Έχουμε ξεκινήσει μια ομάδα εργασία σε τακτικό επίπεδο όπου συμμετέχουν η Uniformed, η Frontex και οι Ιταλικές ναυτικές επιχειρήσεις. Συζητάμε. Έχουμε την ίδια ναυτική εικόνα. Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που λειτουργεί πολύ καλά. Ευχαριστώ. We know that there are... Γνωρίζουμε ότι εδώ έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελε κάποιος να συμμετάσχει, αλλά πολύ σύντομα δυστυχώς, ε, ώστε να μας πείτε αν υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων οδών. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ωραία, συγγνώμη. Ωραία, η Frontex πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τις εναλλακτικές οδούς μετανάστευσης, σύμφωνα με τις αναλύσεις της Frontex, μπορούμε να πούμε ότι προς το παρόν, οι μετανάστες που έχουν παραμείνει αποκλεισμένοι στην Ελλάδα αναμένουν στην Ελλάδα είναι κάπου μεταξύ 50 με 70 χιλιάδες οι μετανάστες που έχουν μείνει μπλοκαρισμένοι στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι ο αριθμός των αφήξεων τώρα έχει μειωθεί κατακόρυφα. Ε, των αφήξεων μιλάμε από Τουρκία προς Ελλάδα έχουμε κατά όρο 100 μετανάστες συμμερισίως. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί μετανάστες περιμένουν επίσης και στην Τουρκία. Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις που να μας λένε ότι υπάρχει μετατόπιση της δραστηριότητας από την Τουρκία στη Λιβύη. Ωστόσο υπάρχει αύξηση των αφήξεων από τη Λιβύη στην Ιταλία, αλλά ε, αυτοί οι μετανάστες προερχόνται από άλλη πηγή ε, προερχόνται λόγω εξελίξεων στην Αφρικανική Ήπειρο, αλλά δεν είναι οι ίδιοι όπως αυτούς που έρχονταν από την Τουρκία. Η Frontex το παρακολουθεί και είμαστε έτοιμοι να ε, ξεκινήσουμε νέε δραστηριότητε αν χρειαστεί. Όσον αφορά τι εναλλακτικέ οδού ε, από την Τουρκία μέσω του Ευξηνού Πόντου, ενδεχομένω προ τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, μόνο με μονομένε περιπτώσει μέχρι στιγμή. Δεν αποτελεί λοιπόν οδό. Όσον αφορά πιθανές εναλλακτικές οδούς ε, μέσω της Αλβανίας, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι ακόμη, πέραν κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων που κινούνται από τη δυτική ακτή της Ελλάδας προ, απευθείας προς την Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, σε συμφωνία με τις Ιταλικές Αρχές, η Frontex έχει επεκτείνει τον χώρο των επιχειρήσεων και στην Αδριατική, ώστε να παρακολουθεί με ενέργεια μέσα πιθανές διελεύσεις από την Αλβανία προς την Ιταλία ή από το Μαυροβούνιο προς την Ιταλία. Μέχρι στιγμής όμως η κατάσταση φαίνεται να έχει παραμείνει στάσιμη. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν προς τη Frontex. Όσον αφορά τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ευρωπόλ και Frontex, όσον αφορά την ιστορική ασφάλεια, στην εντολή που πρότεινε η Κομισιόν αλλά και στο κεκτημένο Σέγγεν αναφέρεται ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ιστορικής ασφάλειας. Όπως καταλαβαίνω εγώ λοιπόν, τα εξωτερικά σύνορα είναι ένα φίλτρο όπου ελέγχονται οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα πριν εισέλθουν ή εξέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως ε, Frontex ε, αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στην ανείχνευση πιθανών απειλών. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ εμάς και της Ευρωπόλου στα hot spot στην Κατάνια. Αναπτύξαμε πλέον ε, το έργο Πέτρα, όπου η Frontex ενημερώνει ε, ε, ε, συνομιλαμβάνει προφορίες από τους μετανάστες, συλλέγει δεδομένα για πιθανά εγκληματικά δίκτυα και διακινητές. Συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα διαβιβάζουμε στην Ευρωπόλ και στις εθνικές αρχές, σε αυτή την περίπτωση στις Ιταλικές αρχές και μετά από την αστυνομία και στις δικαστικές αρχές να προχωρήσουν σε έρευνα των υποθέσεων αυτών. Ένα άλλο παράδειγμα συνεργασίας που έχουμε είναι στα ελληνικά hotspot παρότι δεν έχουμε κάποιο νομικό πλαίσιο που να μας επιτρέπει την πρόσβαση στο SIS. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπόλ χρησιμοποιεί το εθνικό προφίλ των συνδροφυλακών που υπάρχουν εκεί για να ελέγχει τις ταυτότητες στο Schengen Information System. Οπότε υποστηρίζουμε την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, διότι μιλάμε για ε, υπέργο αριθμό ε, ανθρώπων που πρέπει να ελεγχθούν. Επίσης έχουμε τώρα και τους συναδέλφους της Ευρωπόλ τόπου, οι οποίοι ερευνούν ύποπτε περιπτώσει που έχει ανοιχνεύσει η Frontex και έχει διαβιβάσει στην Ευρωπόλ και έτσι εκεί η Ευρωπόλ μετά χρησιμοποιεί τις δικέ της ειδικευμένε, α πούμε βάσει δεδομένων. Για μένα λοιπόν οι εξελίξεις στα hot spot τη Ιταλία και τη Ελλάδα. δείχνουν τι μορφή θα μπορούσε να έχει ευρύτερη κλιμακά η συνεργασία μεταξύ Frontex και Ευρωπόλ όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια. Και δείχνουν και ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ε, οργανισμών μας και των αποστολών μας. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει επαρκή συμπληρωματικότητα, αρκετή δουλειά για όλους ε, και φυσικά βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα. Τώρα, όσον αφορά την ακτοφυλακή και την πρόταση της Κομισιόν, η άποψή μου για την ανάπτυξη της ακτοφυλακής ε, στο πλαίσιο της Frontex είναι ότι η ακτοφυλακή σε κάποιο βαθμό είναι η θαλάσσια συνοριοφυλακή. Είναι ο θαλάσσιος οργανισμός επιβολής του νόμου και φυσικά έχει το καθήκον ε, έρευνας και διάσωσης ε, και φυσικά η Frontex ασχολείται με όλα αυτά, οπότε αποτελεί καλή εξέλιξη αλλά και φυσιολογική εξέλιξη. Το ότι σε κάποιο βαθμό η Frontex αποκτά αρμοδιότητες στο πεδίο της ακτοφυλακής. Αλλά πρέπει να πω ότι η ακτοφυλακή όσον αφορά την υλοποίηση του ε, κώδικα σύνορων Σέγγεν, ε, όσον αφορά την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τις αρχές εμβολής του νόμου, τα τελωνία και φυσικά και για την έρευνα και διάσωση. Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την περιβολητική προστασία, ε, αυτά είναι αρμοδιότητες άλλων οργανισμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε με την ΕΜΣΑ και την ΕΦΚΑ, αλλά ε, αποτελούν τελείω διαφορετικέ ε, δραστηριότητε. Ένα περαιτέρω ερώτημα αφορούσε το τι θα γίνει. Όχι, όχι, νομίζω τα κάλυψα όλα. Ναι, ναι, συγγνώμη, γιατί έχουμε άλλους τρεις ομιλητές οι οποίοι περιμένουν αδειμόνως. Και καθυστερούμε ιδιαίτερα σε σχέση με τον χρόνο. Θα ήθελα να μην πιέσω τους δύο ομιλητές, αλλά παρακαλώ παραμείνετε μέσα στα δύο ή τρία λεπτά το πολύ. Ναι, και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, λέει ο κύριο Μαρτίνου. Προσπαθώ να ομαδοποιήσω τα διάφορα ερωτήματα που έθεσαν οι αξιοτιμικοί βουλευτέ. Δεν ξέρω. Υπήρξε το θέμα τη ε, διαλειτουργικότητα των δεδομένων. Αυτό είναι κέριο ερώτημα. Το θέμα αυτό σημαίνει ότι πρέπει καταρχήν να χρησιμοποιούμε πλήρω αυτά που έχουμε στη διαθέσή μας. Δεν γίνεται ακόμα κάτι τέτοιο. Όλα αυτά που είναι διαθέσιμα δεν την χάνουν πλήρως εκμετάλλευση. Βέβαια υπάρχουν ε, εμπόθια ε, σε νομικό ή τεχνολογικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και η εντύπωση ότι θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια γιατί υπάρχει μια προστιθέμενη αξία που μπορεί να προέλθει από την εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων. Δεύτερον, πριν από λίγες εβδομάδες ήταν σχεδόν αδιανόητο το σύστημα πληροφόρησης του Σέγγεν θα μπορούσε να συνδέεται με τεχνικά συστήματα, οι τεχνικά συστήματα θα μπορούν να ελέγχουν το ένα το άλλο. Τώρα όμως είμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι απαραίτητο να διασταυρώνται όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί μπορεί πληροφορία για ένα ύποπτο να βρίσκεται σε μια άλλη βάση δεδομένων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Θα πρέπει να φτιάξουμε νέα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Πρέπει να ξεπεράσουμε τεχνικά προβλήματα, αυτό είναι εύκολο. Πρέπει να ξεπεράσουμε και νομικές, νομικές πτυχές, νομικά προβλήματα και υπάρχουν και τα θέματα αυτά, όπως είπε ο κ. Ιέλερ, σε σχέση και με τη μετάφραση. Είναι πολύ σημαντικό για την ταυτότητα ενός ατόμου να έχουμε ένα ενίο τρόπο να ξέρουμε ποιος είναι ποιος, είτε έχει γραφτεί το όνομά του στα μανδαρίνικα ή στα αραβικά. Και ότι δεν θα προέλθει από λόγους μετάφρασης κάποια δυνατότητα διαστόφρασης, στοιχείων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν κάποιο κοινό πρότυπο και θα πρέπει να τυποποιηθούν και οι νέες βάσεις δεδομένων που θα δημιουργηθεί. Αυτό για τη διαλειτουργικότητα, τα hot spots, εκεί πραγματικά η Frontex έπαιξε ένα πολύ σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο, ιδίω για την Ελλάδα και την Ιταλία, υποστήριξε τις αρμόδιες αρχές. Για τη συνεργασία εν Frontex με την Europol, υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαβίβαση προσωπικών στοιχείων Πιστεύω ότι όλα αυτά θα συμπληρωθούν σύντομα. Ήδη τα χρησιμοποιούμε για έρευνες. Τα εμπόδια, ναι βέβαια υπάρχουν ακόμα εμπόδια, υπάρχουν κενά και χαίνοντα χάσματα στην πληροφόρηση γιατί ορισμένα δεδομένα δεν την χάνουν μου. Όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει με το ταχύτερο δυνατό να διαβιβάζονται, να χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων που έχουμε και να μπορούν τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων να χρησιμοποιούνται και από άλλες διοκτικές δυνάμεις. Ε, επίσης το οργανωμένο έγκλημα για μένα είναι πολύ δύσκολο να, να <clears throat> σας πω πόσα χρήματα από τα έσοδα έχουν να κάνουν και με τρομοκρατία. Έχουμε την περίπτωση αυτών των δραστών στα στην ε, τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στο Παρίσι που ήρθαν ως <clears throat> μεταμφιεσμένοι πρόσφυγες. Επίσης έχουμε την παρουσία του Ισλαμικού κρατού στη Λιβύη που διευκολύνει την ε, διακίνηση ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουν χρήματα με αυτές τις δραστηριότητες. Δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε σαφείς πληροφορίε από τη Βόρεια Αφρική, δεν έχουμε συμφωνίες ακόμα Έχουμε όμως συμφωνίες με την Ιντερπολ, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Με... Το θέμα είναι να μπορέσουμε να έχουμε πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν νομίμως και οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της ασφαλείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιο άλλο ερώτημα που ετέθη για την ε, εισαγωγή λαστιγένιων σκαφών. Εάν κάτι είναι αντικείμενο υποψία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικέ ε, ενέργειε, μπορεί να κατασχεθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε πληροφόρηση ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αγαθά για την διαξαγωγή εγκλημάτων, αδικημάτων και αντιμετωπίστηκαν ως απλά αθώα εμπορικά αγαθά. Ήρθαν λοιπόν αυτά τα πλοία από την Κίνα ώστε να πάνε στη Λιβύη, αν ξέρουμε κάτι τέτοιο, αν έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες εγκαίρως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατάσχεση αυτών των αγαθών. Δίνω και πάλι το λόγο στον πρόεδρο, αν θέλει κάτι το οποίο ξέχασα μπορεί σε μια άλλη συνάντηση, σε μια άλλη στιγμή να το καλύψουμε. Ναι, ναι, είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία μπορούν να λεχτούν και χαίρομαι που υπήρξε αυτή η κοινή παρουσία όλων των φορέων γιατί μπορούμε να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες και σας ευχαριστώ. Και τέλος η κυρία Πρέσβης. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Τρία ερωτήματα απευθύνονται σε μένα. Για το αν υπάρχουν πλοία του ΝΑΤΟ στην ε, περίμετρο της Λέσβου και σε διεθνή ύδατα. Η απάντηση είναι ναι. Θέλω να σχολιάσω για τη συμφωνία ε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας, αλλά δεν δική μου αρμοδιότητα, και επίση για την συμμετοχή τη πολιτική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Βέβαια, αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΝΑΤΟ και αυτή είναι η πιο πολιτική ενέργεια, αλλά υπάρχει και μια σημαντική επιτροπή που λέγεται Operational Policy Committee, Λειτουργική Επιτροπή πολιτική, η οποία πρέπει να τα εγκρίνει όλα αυτά. Επίση για τη σχέση του ΝΑΤΟ και τη EU Ναβφόρτ και του ΝΑΤΟ. Εγώ σας παραπέμπω σε αυτά που είπε ο κ. Κατεντίνο. Υπάρχει μια άτυπη αλλά πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Σε πρακτικό επίπεδο γίνεται συνεργασία. Κατά την άποψή μας λοιπόν λειτουργεί πολύ καλά και η ελπίδα μας είναι ότι η διάδραση αυτή και η συνεργασία άτυπη, έντυπη ή επίσημη θα μπορέσει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν τις βέλτιστες αυτές τις πρακτικές που θέτουμε σε εφαρμογή με την εμπειρία μας στο Αιγαίο. Το επόμενο ερώτημα, τι γίνεται στους μετανάστες οι οποίοι διασώζονται. Πρώτα απ' όλα, αν τους διασώσει το ΝΑΤΟ σε τουρκικά νερά. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, είναι ακόμα μια υποθετική περίπτωση, ένα υποθετικό σενάριο. Αν όμως υπάρξει μια τέτοια περίπτωση που διασώζονται άτομα στα τουρκικά χωρικά ύδατα θα πρέπει καταρχήν να επιστραφούν στα, στην Τουρκία αλλά ο κυβερνήτης του πλοίου που θα κάνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να σεβαστεί το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Επομένως πρέπει να γίνει μια κατά περίπτωση αξιολόγηση για το τι πρέπει να γίνει αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις έχουμε ψάφσει την επιφάνεια της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Χαίρομαι, χαίρομαι που το κάνουμε αυτό και ξαναδίνω το λόγο στην Συμπρόεδρο Άννα Φωτίγα. Εγώ πρέπει να φύγω στις 5 βέβαια και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση αυτή και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πολυαρίθμος ήταν παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση. Ξέρω ότι είχαμε πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε σήμερα το πρωί και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας και να παρακαλέσω την γραμματεία να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να περάσουμε στο επόμενο πάνελ, το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα στις ε, έρευνες ε, για τους διακινητές και τις διώξεις εις βάρος τους. Σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε τους επόμενους ομιλητές μας. Ευχαριστώ.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 Okay, Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας, που είναι το δεύτερο πάνελ. Εδώ είναι πιο πολύ τα θέματα της ε, αποφασίσαμε να δείξουμε και τη θαυμάσια συνεργασία μεταξύ τη Σέντε και τη ΛΥΜΠΕ και το επόμενο πάνελ όπου προεδρεύω εγώ είναι πιο πολύ στις αρμοδιότητες της ΛΥΜΠΕ. Το θέμα μας είναι ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων. Σας παρακαλώ. αυτοί που αποχωρούν μήπως μπορούν να το πράξουν ηρέμως και ησύχως ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Θέλουμε λοιπόν το σεβασμό των ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, ενώ συγχρόνως θέλουμε να γίνεται η δίωξη των διακινητών. Έχω λοιπόν την τιμή να σας παρουσιάσω τους τρεις διακεκριμένα. Ε, τα τρία μέλη του πάνελ έχουμε καταρχήν τον ε, δημόσιο, τον εισαγγελέα του, του της του Παλέμου, τον κύριο Μαρίτσιο Σκάλια. Χαίρομαστε πολύ για την παρουσία του. Μετά έχουμε το γερμανό εθνικό εκπρόσωπο στο σύστημα Eurojust, τον κύριο Klaus Μάιερ Κάμπριμ. Και τρίτο, είναι ο αντιπλήρχος Ολιβιέ Ντασίλβα, ο πλήρχος μάλλον Ολιβιέ Ντασίλβα, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος στην UNAFOR Σομαλία με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ε, διερεύνηση αδικημάτων. Εκεί πέρα πρόκειται για πειρατές. Αλλά έχουμε πολύ καλές εμπειρίες ήδη σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Αταλάντα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που αφορά περισσότερο την ΣΕΔ. Περιορισμένου όντως του χρόνου θα ήθελα να δώσω αμέσως και ακαριέως τον λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Σκάλια. Έχετε το λόγο. Ε, ναι, ευχαριστώ. Η ομιλία μου αφορά τις ε, τρέχουσες διαδικασίες ε, στην εισαγγελία του Παλέρμο, όπου ονομάζονται Γκλάκο 1 και Γκλάκο 2 κωδικοποιημένα. το ότι μίλησα μετά από τον εκπρόσωπο του ναυτικού της Ευρωπόλ και της Frontex έχει νόημα διότι η έρευνα της εισαγγελίας του Παλέρμου και των υπολείπων Ιταλικών εισαγγελιών έρχονται, είναι το επόμενο βήμα και συγκεντρώνουν ουσιαστικά και επεξεργάζονται αυτά τα στοιχεία. Στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου ήθελα να σας περιγράψω πώς ξεκινούν αυτές οι διαδικασίες ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και ποιες είναι οι προτάσεις μας για λύσεις. Σε αυτές τις διαδικασίες ε, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ στενή σύνδεση, όπως μαθαίνουμε από τους ανθρώπους ε, και τους τρόπους που διακινούνται στη Βόρεια Αφρική ε, με τους διακινητές ανθρώπων. Υπάρχει επαφή με άλλους οργανισμούς της Ιταλίας που υποδέχονται τους μετανάστες και μετά τους μεταφέρουν στις χώρες της Κεντρικής και Βορειάς Ευρώπης. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 2013 όταν βρήκαμε έναν από τους διακινητές ε, ανθρώπων, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για το τραγικό ναυαγείο της 3ης ε, Οκτωβρίου του 2013, όπου έχασαν τη ζωή τους 366 άτομα έξω από τη Λαμπεντούζα. Ο διακινητής αυτός ε, συλλήφθηκε μετά από ένα μήνα στην Ιταλία και καταδικάστηκε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σε 30 ε, κονταετή φυλάκιση. Αυτό οδήγησε σε έρευνες με στόχο το να μην περιοριστούμε στη σύλληψη των διακινητών. Συχνά όταν μιλάμε για διακινητές ε, αναφερόμαστε στους πλοηγούς των σκαφών. Μέσω λοιπόν των πληροφοριών και των δηλώσεων των μεταναστών και μέσω των τηλεφωνικών υποκλοπών έχουμε καταφέρει να αναπαραγαγούμε την αλυσίδα αυτών των δραστηριοτήτων που ξεκινούν από τη Βόρεια Αφρική και μέσω των τηλεφωνικών υποκλοπών καταφέραμε να βρούμε τρεις από τους βασικούς διακινητές ε, ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στη Λιβύη και λειτουργούν από εκεί. Είναι ένας Σουδανός, ε, ένας Ερυθρέος ε, ένας και ένας Αιθίωπας ξέρουμε τα ονόματα και τα επώνυμά τους και έχουμε εκδώσει ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Έχουμε επεκτείνει τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο, αλλά όπως κατέβεται αυτή τη στιγμή το να συλλάβουμε κάποιον στη Λιβύη είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Ε, είναι ε, αυτές οι λήψεις εξαιρετικά δραματικές γιατί Ε, όταν ε, συλλέξαμε τις πληροφορίες για το θάνατο αυτών των 366 ανθρώπων, αντιληφθήκαμε την αδιαφορία αυτών των ανθρώπων ε, για την τύχη αυτών των μεταναστών. Η μόνη τους ανησυχία, το μόνο που τους απασχολεί είναι να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και το δικό τους ε, στάτους να μην αλλάξει για, από αυτό το απλό για αυτούς περιστατικό Στην επιχείρηση Γκλαουκό 1 είχαμε ήδη τις πρωτοβάθμιες ε, καταδίκες των ατόμων ε, που στην Ιταλία συνεργάζονται με τους ε, Λίβιους διακινητές και για τη μεταφορά των μεταναστών στην Κεντρική και Βορεια Ευρώπη στην επιχείρηση Γκλαουκό 2 έχουμε 24 ανθρώπους οι οποίοι έσταλεσαν στη δικαιοσύνη και στην πλειοψηφία τους, για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν προφυλακιστεί. Καταφέραμε να, να, δούμε... να φτιάξουμε και την εικόνα του τρόπου ε, λειτουργίας όλων, όλης αυτής της αλυσίδας. Πρόκειται για δραστηριότητες ε, ε, που προσφέρουν τεράστια κέρδη. Ουσιαστικά κάποιος που προέρχεται από τη Σομαλία, την Ερυθρέα ή το Σουδάν πληρώνει περίπου 5.000 ευρώ για να φτάσει μέχρι τη Λιβύη. Εάν ξεφύγει από ε, τις απαγωγές ε, στο Σουδάν και στο κέντρο της Λιβύης ε, και αφού φτάσει στη Λιβύα για να περάσει στην Ιταλία πρέπει να καταβάλει επιπλέον 1600 δολάρια και μετά το τελικό σκέλος ταξιδιού από την Σικελία μέχρι το κέντρο της Ιταλίας ε, κοστίζει κάπου 200 με 400 ευρώ και μετά για να πάει προς τις χώρες κεντρικής και βορειάς Ευρώπης πρέπει να καταβάλει μεταξύ 1000 και 1200 ευρώ. Εάν το πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό των αφήξεων Σομαλών, Ερυθρέων και Σουδανών στην Ιταλία από το 2014 37.177 άτομα και 49.000, ε, ε, λίγο παραπάνω από 49.000 άτομα το 2015. Μιλάμε για τεράστια ποσά, διότι ξέρετε και οι δαπάνε των οργανισμών αυτών είναι απειροελάχιστε. Ε, σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται πολλές φορές, ε, ε, ε, φορτηγάκια ή χώροι όπου φυλάσσονται οι απαχθέντες μετανάστες. Αυτή δεν είναι η μόνη δυσκολία. μονη δυσκολια προκειται για πολλούς, πολυάριθμους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευέλικτοι. Όλα αυτά που σας λέω έχουν επιβεβαιωθεί ως γεγονότα προσαρμόζονται οι οργανισμοί αυτοί στις πολιτικές συνθήκες. Αν υποθέσουμε ότι στην Αίγυπτο τραβήξουν την προσοχή των αστυνομικών αρχών, τότε οι οργανώσεις, όπως έχει συμβεί και συμβαίνει ακόμη, μεταφέρονται στη Λιβύη. Πρόκειται για οργανώσεις εξαιρετικά ευέλικτες. Όταν εμείς ως εισαγγελία του Παλέρμο το διαπιστώνουμε αυτό, ε, ε, έχουμε κάνει το ίδιο και με μαφιόζους. Ε, όταν τους συλλαμβάνουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή δημιουργούμε δυσκολίες στις μαφιόκες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά στην περίπτωση αυτή των διακινητών δεν συμβαίνει το ίδιο, διότι υπάρχει τεράστια προσφορά και πάρα πολλοί οργανισμοί. Εξαιρετικά ευέλικτο όπως είπαμε, διότι όταν εμείς αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε τους διακινητές, τους πλοηγούς, περίπου 100 πέρυσι, οι διακινητές κατάλαβαν ότι ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και άρχισαν να συνοδεύουν τον κόσμο μέχρι τα όρια των ε, διεθνών υδάτων στα ανοιχτά της ε, ε, Λιβικής ακτής και μετά γυρνούσαν πίσω καλώντας σε βοήθεια μέσω δορυφορικών μέσων. Μια άλλη δυσκολία και το αρχίζουμε να διαβλέπουμε το πρόβλημα της διεθνούς συνεργασίας. Η άλλη δυσκολία λοιπόν είναι ότι τα τόσο υψηλά χρηματικά ποσά δεν είναι ανοιχνεύσιμα, διότι η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιούν εγκληματικές οργανώσεις, ε, η μέθοδος Άβαλα, δεν έχει κανένα κόστος. Διότι δεν εμπλέκονται τράπεζες. Τα χρήματα λοιπόν φτάνουν σε περιοχέ, ή ξεκινώ περιοχέ που δεν υπάρχουν τράπεζε. Πολύ αποτελεσματικά δηλαδή και δεν είναι ανιχνεύσιμα αυτά τα ποσά. Μια άλλη δυσκολία αφορά το γεγονό ότι πρόκειται για διακρατικού οργανισμού, διεθνικού οργανισμού. Οπότε είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ διαφόρων αστυνομικών αρχών και διαφόρων δικαστικών αρχών. Φανταστείτε ότι η πρώτη επαφή του μετανάστη με την εγκληματική οργάνωση ε, γίνεται με κάποιον στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή ο συγγενής του μετανάστη πληρώνει και μετά έχουμε τη μεταφορά από την Ερυθρέα στη Λιβύη, στην Ιταλία, στις χώρες της Βορειάς Ευρώπης. Η καθεμία από αυτές τις φάσεις κάποιοι ε, διακινητές ε, συμμετέχουν σε αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές είναι οι κύριες δυσκολίες. Τι προτάσεις έχουμε ως λύσεις. Κάποιες δραστηριότητες συντονισμού σίγουρα που πρέπει να ξεκινούν ε, αυτή τη στιγμή στα πλοία περισυλλέγουν τα σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες σε διεθνή ύδατα. Μία άμεση κοινοποίηση του συμβάντο στην εισαγγελία της Ιταλικής Δημοκρατίας βοηθά το συντονισμό της έρευνα. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης των αξιωματικών συνδέσμων που βρίσκονται πάνω στα πλοία οι οποίοι μπορεί ήδη να μας δώσουν κάποιες ενδείξεις ε, για το ποιο ε, επιβαίνουν στο σκάφος ε, είναι διατεθειμένος να μας δώσει πληροφορίες για να βρούμε τους διακινητές. Μπορεί δηλαδή να μας δώσει και το τηλέφωνο ενός μετανάστη. Αυτό είναι κάτι πολύ απαραίτητο Επίσης είναι απαραίτητες ε, οι, φω... φωτογραφίες και τα βίντεο των σκαφών ώστε όταν το σκάφος αυτό φτάσει προς το πλοίο που πραγματοποιεί τη διάσωση να μπορούμε να δούμε ποιος δεν είναι πια πάνω ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον διακίνητη και να εντοπίσουμε και την κατάσταση του σκάφους. που σε μερικές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Γιατί σε περιπτώσεις ε, που έχουμε νεκρούς ε, έχουμε το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Φυσικά όταν κάποιος βάζει πάνω σε ένα σκάφος ε, που χωράει 50 άτομα 500 είναι προφανώς ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω κυρικών συνθήκων ή λόγω άλλων προβλημάτων να υπάρξουν νεκροί. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό και θα μιλήσει για αυτό σίγουρα το μέλος της Eurojust είναι ότι αυτή η ροή πληροφοριών που εμείς έχουμε αποκτήσει μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών, μέσω ερευνών και ανακρίσεων ε, όλες αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε διαθέσει μέσω της Eurojust και στις άλλες εισαγγελίες ε, και αστυνομικές αρχές ε, στην Ευρώπη. Αυτό πιστεύω υπήρξε και το πιο ωφέλιμο και ακολούθησε και συνεδρίαση συντονισμού με χώρες διάφορες. Συχνά έχουν έρθει αστυνομικές αρχές εισαγγελίες στο Παλέρμο και πετύχαμε καλά αποτελέσματα, πολύ τακτικά, διότι καταφέραμε να βρούμε ονόματα και επώνυμα των διακινητών ή τι γυναίκε του. Η γυναίκα ενό, για παράδειγμα, βρισκόταν ε, στη Σουηδία. Είχε ένα προφίλ στο Facebook και εμεί καταφέρουμε μέσω τη συνεργασία με τη Σουηδική Αστυνομία να βρούμε τη φωτογραφία αυτού του ανθρώπου και την ημερομηνία γέννησή του. Οπότε να εκδώσουμε ένα ευρωπαϊκό μας σύλληψη. Αυτή η συνεργασία είναι απολύτω απαραίτητη. Διότι οι οργανώσει αυτέ, όπω είπαμε, είναι διεθνικέ. Υπάρχουν επαφές και έχουμε αποδείξεις ε, μεταξύ οργανώσεων στη Λιβύη, με οργανώσεις στην Ιταλία και με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στην Κεντρική και στη Βορεια Ευρώπη. Είναι λοιπόν σαφές ότι όσο καλή και αν είναι μια αστυνομική επιχείρηση, αν δεν υπάρχει συντονισμός ε, με τις υπόλοιπες χώρες ε, και συλλαμβάνεται ένας διακινητής, ο οποίο μεταφέρει 5-6 άτομα στη Βόρεια Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι άσχημο, αλλά είναι, τα αποτελέσματα είναι καλύτερο όταν υπάρχει συντονισμό. Όταν καταφέρνουμε να ταυτοποιήσουμε τους διακινητές, να βρούμε του αριθμού τηλεφώνων τους, αν καταφέρουμε να κάνουμε τηλεφωνικές υποκλοπέ και να προσδιορίσουμε τα άτομα υποδοχής στις διάφορες ε, χώρες της Ευρώπης και να προσδιορίσουμε και τις επαφές που έχουν με τους διακινητές. Επίσης όλα αυτά μας βοηθούν να ε, εντοπίσουμε τις ε, χρηματικές ροές που αφορούν αυτά τα άτομα στις διάφορες χώρες γιατί πολύ συχνά υπάρχουν χώρες συγκεκριμένη υποδοχή των μεταναστών όπου υπάρχουν και κανονικές και ε, παράνομες δραστηριότητες ε, και όπου υπάρχουν ε, κινήσεις χρημάτων μεγάλων διαστάσεων. Αυτό βέβαια αφορά τις τρέχουσες έρευνες και είναι κάτι απολύτως απαραίτητο διότι όπως είπα στις χώρες της Βορειοαφρικής εμείς έχουμε εντοπίσει κάποιους διακινητές. Η ταυτοποίηση τους ε, και η μετακίνησή τους σε χώρες με τις οποίες εμείς έχουμε ε, συμφωνίες απέλασης είναι κάτι επιθυμητό και θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη ε, των εν λόγω ανθρώπων. Πιστεύω ότι υπήρξα αρκετά συνοπτικός. Είχα να πω πολλά ακόμα, αλλά ουσιαστικά ήθελα να σας παρουσιάσω πώς γίνονται οι έρευνες, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες ήταν οι λύσεις. Ε, αυτά και σας παρουσίασα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαγγελέα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Ακολουθούμε τώρα τον επόμενο εμπειρογνώμονα για τα θέματα λίμπε είναι ο κύριος Κλάους Μάιερ Κάμπρι που είναι ο Γερμανός Εθνικός Εκπρόσωπος στην Eurojust. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορώ να συνδεθώ αμέσως με αυτά που είπε ο συνάδελφος από το Παλέρμο. Είναι κέρια η συνεργασία και ο συντονισμός. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Eurojust το 2002 και τότε ήμουνα νέος. Ήμουνα νέαρος νομικός σύμβουλος και είχαμε τότε το πρώτο, το πρώτο μου έργο ήταν το νομικό πλαίσιο της Eurojust. Είμαι λοιπόν πολύ γέρο με τη Eurojust. Και η Eurojust έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις εθνικές εισαγγελικές αρχές για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις όπου ένας εγκληματικός οργανός οργανισμός βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες. Πρόκειται λοιπόν για τον αγώνα κατά του διαμεθοριακού εγκλήματος, αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε ιδίως σε περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών, λα, λαθρεμπορίας μεταναστών, είναι να υπάρξει μια ουσιαστική ε, αντιμετώπιση των διακινητών. Αυτό το οποίο είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα και το τονίζει και η ακρόασή σας είναι να έχουμε την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Αλλά οποιαδήποτε δίωξη πρέπει να γίνει επί τη βάση του κράτους δικαίου. Δεν μπορούμε να αναστείλουμε το κράτος δικαίου επειδή τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μεγάλα. Μια περίπτωση τώρα να σας αναφέρω όπου ο ρόλος της Euro Just ήρθε να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση. Είναι η περίπτωση Λόρι, όπως είναι γνωστή. Η, μάλλον η περίπτωση του φορτηγού. 71 ε, μετανάστες πέρασαν σε ένα φορτηγό μέσα τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και έχασαν τη ζωή τους στην ε, Ουγγαρία, αλλά τους βρήκαν στην Αυστρία. και υπήρχαν και κάποιες ε, διασυνδέσεις με τη Γερμανία, οπότε εμπλέκονται τέσσερα κράτη-μέλη στην περίπτωση αυτή. Πρέπει να φέρει κανείς από κοινού τις ε, διοκτικές και εισαγγελικέ αρχές των τεσσάρων χωρών για να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό έγινε λίγο μετά από την ανακάλυψη των 71 νεκρών μεταναστών στην Αυστρία τον Αύγουστο του 2015 ακολούθησε διαδικασία στα, στο αρχηγείο της Eurojust και στην δικαστήριο της Χάγης, γιατί εκεί πρέπει να προκύψει μια συμφωνία για το ποιος θα πρέπει να κάνει την ε, διαδικασία έρευνας και ανάκρισης. Οι Αυστριακοί εκεί πέρα ε, είπαν ότι αυτοί δεν θα ασχοληθούν και το έδωσαν στην Ουγγαρία. Υπήρχαν όμως και συνδέσεις με άλλες περιπτώσεις. Υπήρχε το ερώτημα του πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει τη συνεργασία με κοινέ ομάδες έρευνας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται, γιατί είπαν οι Γερμανοί ότι όσες πληροφορίες έχουμε μπορούμε να τις δώσουμε αμέσως στους Ούγγρους. Γιατί οι Ούγγροι χρειαζόταν σε αυτές τις πληροφορίες. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λοιπόν βρέθηκαν άλλες έξι περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών που συνδεόντουσαν με την προηγούμενη και πρέπει να ληφθούν και αυτές οι υπόψει. Αυτό όμω είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συνενώνουν τις προσπάθειές τους, να βρίσκουν μια κατανομή έργου, να βρίσκουν πώς μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες και να τις εκμεταλλεύονται. Η Eurojust σε τέτοιες περιπτώσεις έχει τρία κύρια εργαλεία. Το πρώτο το έχω αναφέρει προηγουμένως, είναι οι συναντήσεις συντονισμού, όταν όλοι οι εθνικοί εμπλεκόμενοι εισαγγελείς έρχονται σε επαφή και συνεννοούνται μεταξύ τους. Το δεύτερο είναι τα κέντρα συντονισμού που οργανώνουν κοινέ δράσεις. Δηλαδή στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται συγχρόνως συλλήψεις, κατασχέσεις και αυτό έχει οργανωθεί από την Eurojust. Και επίση έχουμε και τις κοινέ ομάδες ανάκρισης όπου βασίζονται σε μια συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών για το πώς θα γίνουν κοινέ έρευνες και ανακρίσεις για την διαλεύκανση αδικημάτων. Και εκεί το πλεονέκτημα είναι ότι, ότι βάσει αυτών των συνθήκων μπορεί κανείς να διαβιβάσει πληροφορίες χωρίς να υπάρξουν επίσημες αιτήσει για αρρωγή, δηλαδή να ζητήσει μια χώρα μια άλλη για νομική αρρωγή. Όλο αυτό επιταχύνει τη διαδικασία. Κάτι άλλο το οποίο κάνουμε επίσης είναι ότι δίνουμε στους εμπλεκόμενους εισαγγελείς εργαλεία για να κάνουν με καλύτερο τρόπο την εργασία τους. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που βρίσκονται μέσα στην νομολογία μας. Η νομολογία λοιπόν αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι από τις εισαγγελικέ αρχές. Είναι μια ανατροφοδότηση σε πληροφορία περί του πρακτέου. Αν παραγωγός χάρη αν έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών και έχετε βρει τον καλύτερο τρόπο να γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι μια βέλτιστη πρακτική. Όλα αυτά μπορούμε να τα δώσουμε στις διάφορες εισαγγελικέ αρχές, που, ιδίως αυτές που το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα για πρώτη φορά και έτσι έχουν ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να τους δώσει κατεύθυνση. Αυτό είναι έμεση λειτουργική συνεργασία και ιδίως σε περιπτώσεις μετανάστευσης είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η συνεργασία μέσω της Eurojust. Πάνω από 50% έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται. Οι συναντήσεις συντονισμού έχουν αυξηθεί κατά 50% το 2015 του 2016 και αυτή είναι μια συνεχιζόμενη τάση το 2016. Δεν υπάρχει λοιπόν χαλάρωση προσπαθειών εδώ. Τι έχει κάνει τώρα η Eurojust για να αυξήσει την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών διακίνησης μεταναστών, όπως είπαμε προηγουμένως. Συνεργαζόμαστε με όλους τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, διαμοιραζόμαστε πληροφορίες και βοηθούμε ο ένας τον άλλο. Γύρω just είναι παρούσα στα hot spots. Τα hot spots είναι πολύ σημαντικά γιατί αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν πρόκειται μονάχα για την καταγραφή των προσφύγων που είναι το πρώτο μέλημα, αλλά είναι και το πρώτο σημείο εισόδου όπου μπορείτε να πάτε πληροφορίες για τη διακίνηση, μπορούν οι μετανάστες να σας πούν για αυτήν την ε, μορφή διακίνησης. Υπάρχουν πολλές φορές και ελάσσονες διακινητές οι οποίοι μπορούν να συλληφθούν παρόντες. Όλα αυτά είναι πληροφορίες από πρώτο χέρι που μπορούν να συλλεγούν πολύ γρήγορα και μετά πρέπει να δοθούν στην συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη. Δεν πρόκειται μονάχα λοιπόν για την Ελλάδα και την Ιταλία, μπορούν να πληροφορηθούν και άλλα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να διαβιβάσουμε αυτές τις γνώσεις που αποκτούμε σε όλους τους άλλους και εκεί βοηθάει η Eurojust. Όπως και η Europol, Έχουμε δημιουργήσει θεματικές ομάδες. Η Europol τα ονομάζουμε κέντρα. εμείς τα, οργάνωτα λέμε ομάδες ή θεματικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα θέματα των μεταναστών και εδώ χρησιμοποιούμε τις γνώσεις που μπορούμε να συλλέξουμε και τις ε, διαβιβάζουμε στις υπηρεσίες των εισαγγελιών που τις χρειάζονται. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι μαζί με τις κοινέ ομάδες έρευνας και ανάκρισης δημιουργούμε ένα κοινό υπόδειγμα για αυτές τις περιπτώσεις. Αν λοιπόν τα εθνικά εισαγγελικά γραφεία θέλουν να δημιουργήσουν κοινέ ομάδες έρευνας και ανάκρισης έχουν και ένα οδηγό που τους λέει πως μπορεί να γίνει αυτό πολύ γρήγορα αυτό. Αναφέρθηκε προηγουμένω από τον κύριο Έλερ στο θέμα της μετάφρασης ή τουλάχιστον σε ερωτήματα στο πρότυνελ και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές οι μετανάστες έρχονται από περιοχές εκτός της Ευρώπης όπου ομιλούνται σπάνιες διάλεκτοι. Άμα κάνετε τηλεφωνικές ε, υποκλοπές. Χρησιμοποιούν μια αργό, μια παράξενη γλώσσα οι διακινητές με τους μετανάστες. Πολύ σπάνια βρίσκεται αξιόπιστος μεταφραστές για αυτές τις γλώσσες. Δεύτερον, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των τηλεφωνικών υποκλοπών που δημιουργεί ένα πρόβλημα. Πολλές φορές λοιπόν είναι τεράστιο το άχθος για τις εθνικές υπηρεσίες να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και η Eurojust μπορεί να βοηθήσει αν είναι μια κατεπίγουσα κατάσταση, αν δεν μπορεί να βρεθεί αξιόπιστος μεταφραστής. Είναι μικρός ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτό και πολλές φορές αυτοί οι μεταφραστές είναι τόσο εμπεπλεγμένοι στην εθνοτική τους ομάδα που δεν πρέπει να τους δώσει κανείς τις αναλύστικες πληροφορίες. Και εδώ τα κονδύλια μας είναι περιορισμένα και θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουν να αυξηθούν τα κονδύλια προ τα κράτη-μέλη, μάλλον των κρατών μελών ή προ την Eurojust για καλύτερη παροχή μετάφραση. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και γενικά εμείς προσπαθούμε να στέσουμε από κοινού τους πόρους μας, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη <clears throat> να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις της ε, παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας των κρατών μελών μπορούμε να ε, διαλευκάνουμε αυτές τις περιπτώσεις πολύ καλύτερα και πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερα εμπόδια από τη με τα φυσιολογικά κανάλια που χρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον πλωτάρχη Ολιβέντε Σίλβερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα. Είμαι νομικός σύμβουλος της Αταλάντα ε, και έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση το 2008 και ο δικός μου ρόλος ε, στην επιχείρηση αυτή είναι νομικός ποια είναι η νομική πτυχή και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Αταλάντα ε, από πολιτικής και νομικής πλευράς σε σχέση με την επιχείρηση Σοφία και ε, τι έχουμε μάθει ε, <clears throat> σχετικά με το τι πρέπει να έχει γίνει από νομικής πλευράς προτού κινητοποιηθεί ένα πολεμικό σκάφος ή αφότου έχουν συλληφθεί ύποπτοι για πειρατεία και θέλουμε να τους διώξουμε ποινικά. Αυτό λοιπόν το legal finish Ε, έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που συλλαμβάνουμε ε, ύποπτους για πειρατεία στη θάλασσα και έχουμε την ευθύνη για αυτούς μέχρι να μεταφερθούν σε κάποιο κράτος μέλος ή αλλού για δίκη. Και ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε επιτυχημένη ποινική δίωξη. Η επιχείρηση Αταλάντα είχε επιτυχία στο θέμα αυτό. 154 υπόπτους ε, έχουμε ε, έχουν προσαχθεί ε, 54 ε, ήταν ύποπτοι, 11 ε, αθώθηκαν και άλλοι περιμένουν ακόμα τη δίκη. Και στην Ιταλία, την Ισπανία και τις Σεϊχέλες και τον Μαυρίκιο είχαμε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό για τους ευρωβουλευτές να καταλάβουν ότι το νομικό πλαίσιο της επιχείρησης Αταλάντα διαφέρει σημαντικά από την επιχείρηση Σοφία. Η πειρατεία είναι θέμα διεθνούς δικαιοδοσίας, το οποίο σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος που θέλει να ασκήσει δίωξη δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει υποστεί ζημιά από ε, την πράξη. Για παράδειγμα, αν έχουμε Σομαλούς ε, πειρατές ε, σε Ινδικό σκάφος, αν του συλλάβουν οι Ισπανοί μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη η Γαλλία, το Ιράν, οποιαδήποτε χώρα, αν θέλει και μπορεί. Η διακίνηση και η εμπορία ανθρώπων διαφέρουν, διότι πρέπει κανείς να δείξει ότι έχει ε, γίνει ζημιά εις βάρος του κράτους μέλους ώστε να έχει επαρκή ε, νομική βάση για να ασκήσει ποινική δίωξη. Η επιχείρηση Αταλάντα επίσης διαφέρει διότι από πολιτικής πλευράς ε, λειτουργούμε εν μέρη υπό τη δικαιοδοσία ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας και είχαμε αρκετά τέτοια ψηφίσματα από το 2008 και μετά σε σχέση με την ε, πειρατεία και Ξεκινήσαμε με τη μεταβατική κυβέρνηση το 2008 και έκτοτε είχαμε πολλές επιστολές από τον πρόεδρο της Σομαλίας όπου καλεί την επιχείρηση Αταλάντα και ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα ε, διαθέσιμα μέσα για να καταπολεμηθεί η πειρατεία. Και μάλιστα και σε φυσικά ύδατα της Σομαλίας ε, αλλά και εις βάρος ε, πολιτών υπηκών της ε, Σομαλίας στη θάλασσα. Η εντολή της επιχείρησης Σοφία είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβέρνηση εθνικής συνένεσης στην Λιβύη. Έτσι λοιπόν είναι αμφίβολο το ότι θα προσκληθούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο εντός της Λιβύης ή εις βάρος υπηκών της Λιβύης στην ανοιχτή θάλασσα και επίσης ε, δεν υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Εφόσον όμως το γνωρίζουμε αυτό, ας προχωρήσω στο τι έχουμε μάθει από την επιχείρηση Αταλάντα και πρωτού ε, κοιτοποιηθεί κάποιο σκάφος και μετά τη σύλληψη προσώπων και την κράτησή τους. Ε, από νομικής πλευράς αποτελείται, ε, είναι απαραίτητη η έγκαιρη ε, συμμετοχή και κινητοποίηση και στις πρώτες μέρες της επιχείρησης αυτής η επιχείρηση Αταλάντα χρησιμοποιούσε την πολιτική capture and release. Συλλαμβάνουμε και απελευθερώνουμε, διότι δεν είχαμε τα νομικά μέσα στη διάθεσή μα ε, που θα μα επιτρέπανε να ασκήσουμε ποινική δίωξη. Και από πλευράς δημοσίων σχέσεων ε, αυτό είναι τρομερό, διότι συλλαμβάνουμε ανθρώπου ε, υπόπτου για πειρατεία, δεν έχουμε όμω τη δυνατότητα να ασκήσουμε ποινική δίωξη. Έτσι λοιπόν ε, στις πρώτες μέρες της επιχείρησης ε, η Αταλάντα ε, είχε συνάψει συμφωνία με την Κένια και είχαμε σύλληψη 79 ατόμων οι οποίοι κρίθηκαν όλοι ένοχοι. Νομίζω οποιοδήποτε εισαγγελέα θα ήταν ικανοποιημένο με τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά το 2010 η Κένια ανακάλεσε τη συμφωνία αυτή και κατόπιν είχαμε συμφωνία με τις Αιχέλες και το Μαυρίκιο για δίκες προσώπων στις χώρες αυτές. Κατά την υπογραφή αυτών των συμφωνιών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να ε, λυθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη ε, και δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύμβαση αυτή ισχύει και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δηλαδή εξωεδαφική ισχύ. Είτε λοιπόν βρισκόμαστε σε διεθνή ύδατα είτε στις ε, εδαφικά ύδατα της Σομαλίας, δεσμευόμαστε ως μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης από ε, τις ε, της, ε, συμφωνίας, της ε, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αυτό έχει να κάνει και με την δίωξη, δηλαδή πώς, τι μεταχείριση θα έχουν οι ύποπτοι για πειρατεία, αλλά έχει να κάνει επίσης και με το χρονοδιάγραμμα και με την επαφή των συγγενών. Επίσης, θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι αυτές οι νομικές ρυθμίσεις ε, σημαίνουν ότι θα κρατούνται άνθρωποι σε πολεμικά ε, πλοία μέχρι να μεταφερθούν είτε σε ε, κάποιο παράκτιο κράτος ή σε άλλο κράτος. Ε, Στι πρώτε 15 μέρε, ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα ασκήσουν ποινική δίωξη. Εάν δεν υπάρχει κράτο μέλο που να θέλει να ασκήσει ποινική δίωξη, ε, δίδονται άλλα 10 άλλες 10 μέρες σε περιφερειακά κράτη, δηλαδή τις σε ή το Μαυρίκιο στη συγκεκριμένη περίπτωση και εάν δεν το θέλουν τότε είμαστε υποχρεωμένοι και πάλι να απελευθερώσουμε τους κρατούμενους. Κατά την διαδικασία για την, ε, για την απόφαση για το ποιος θα ασκήσει δίωξη. Εξετάζουμε δηλαδή πρώτα εάν θέλουν να ασκήσουν ποινική δίωξη τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν τα περιφερειακά κράτη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη και τα περιφερειακά κράτη θα πρέπει να γνωρίζουν περίπου τι ε, τεκμήρια θα έχουμε για να γνωρίζουν εάν θέλουν να ασκήσουν ποινική δίεξη. Ένα πολεμικό σκάφος ε, δεν ε, θα μπορεί να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάποιες ενδείξεις σχετικά με το τι στοιχεία υπάρχουν για να δούνε κατά πόσο θα επιτυχεί η ποινική δίωξη. Τα διάφορα κράτη-μέλη και τα διάφορα περιφερειακά κράτη θα έχουν διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία και αυτό είναι σημαντικό διότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περιφερειακά κράτη να συμμετέχουν στη διαδικασία ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι οι απαιτήσει και τι χρόνος κράτησης ε, των προσώπων αυτών επιτρέπεται. Αλλά ευρωπαϊκά κράτη είχαν προβλήματα όσον αφορά την προσαγωγή των ατόμων εντός 24 ώρου και έπρεπε να πληρώσουν αποζημίωση σε ανθρώπους που εκ των υστέρων κρίθηκαν ένοχοι πειρατεία. Ε, και εδώ λοιπόν εφαρμόζεται η ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όταν ένα πολιτικό πολεμικό σκάφος ε, συλλαμβάνει ύποπτους για πειρατείες, Εάν συμμετέχουν τα πρόσωπα αυτά στην επίθεση, τότε ε, είναι αρκετά εύκολο να ε, αποδείξει κανείς ότι ε, είναι πειρατέ, αλλά εάν δεν πιαστούν επαυτοφόρο εντό αγωγικών, τότε είναι πιο δύσκολο να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία. Όταν τα πρόσωπα αυτά μεταφερθούν στο πολεμικό σκάφο, υπάρχουν χρονικά όρια σχετικά με το πόσο χρόνο μπορούν να διμένουν στο σκάφο αυτό και Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί εάν το πολεμικό σκάφος θα πρέπει να ε, μπει σε λιμάνι, κάτι το οποίο είναι ίσως ε, λιγότερο πρόβλημα στη Μεσόγειο από ότι στο κέρα τη Αφρικής. Ποιο συλλέγει τα ε, στοιχεία στο σκάφος και οι πληροφορίες που θα χρειαστούν για την άσκηση ποινική δίωξη, τα στοιχεία δηλαδή που θα πρέπει να έχει ο εισαγγελέα, μπορεί να μην κρυθούν παραδεκτά στο δικαστήριο και Περιμένουμε έτσι από το στρατό να συλλέξει μαρτυρίες, να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία είτε από τους Σομαλούς είτε ε, από τα ε, φαινόμενα θύματα της υπόθεσης ε, και να τα δώσουν στους εισαγγελείς. Κατόπιν η αστυνομία και η εισαγγελία θα προσέλθουν στο σκάφος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι ο στρατός δεν μπορεί να συλλάβει πρόσωπα. Γενικά δεν έχει την αρμοδιότητα αυτή ο στρατός μπορεί να έχουμε ε, κλιμάκιο της επιβολής ε, του νόμου, όπως ε, συμβαίνει συχνά στην Μεσόγεια, αλλά στις περιπτώσεις συλλήψης στο πλαίσιο της EU e for Atalanta, ε, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτές οι δίκες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και τα στοιχεία που σας έδωσα στην αρχή σχετικά με τους 154 που ε, προσήχθησαν και τους 126 που, ε, κρίθηκαν, που καταδικάστηκαν δείχνει για τι περιπτώσεις μιλάμε. Στις Σεϊχέλες είχαμε μια περίπτωση ε, ε, Ιαπώνων ε, με ελικόπτερο, κάποιων Βρετανών και δεν είναι μια απλή εγχώρια διαδικασία όπου μπορεί κανείς να ζητήσει από κάποιον να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, διότι δεν έχει κάποιο νομικό αποτέλεσμα η κλήση στο δικαστήριο. Πολύ συχνά, αν μιλάμε για μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονται στον Ινδικό ωκεανό, είναι πολύ δύσκολο να τους βρούμε για να δούμε αν είναι διαθέσιμοι για να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου. Οι δικές των πειρατών χρειάζονται χρόνο. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μία μεταφορά στην Γαλλία, αλλά αυτό χρειάστηκε πέντε χρόνια. Οκτώ περιπτώσεις θα ανοίξουν σε διαδικασία έφεσης. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ερώτημα του αν αυτά που έγιναν ήταν αντίθετα με το γαλλικό σύνταγμα και αν διατηρήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα των υπόπτων. Η εμπειρία των κρατών για, που κάνουν αυτές τις δίκες ποικίλει. Κάποιες χώρες είναι ιδιαίτερα πεπειραμένες για το διεθνές δίκαιο, άλλες όχι. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Η UNAFOR Atalanta τα τελευταία 7 χρόνια, χρόνια έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες που έχουν βοηθήσει την δίωξη. Αναφέρθηκε αυτό από τους προηγούμενους ομιλητές. Υπάρχει το θέμα της ε, πληροφόρησης και της ε, συλλογής και θέσης από κοινού στοιχείων. Δεν ε, μπορώ να παραλείψω αυτό το στοιχείο. Έχει η αποστολή αυτή η Αταλάντα <coughs> αξιωματικού συνδέσμους στις Σεχέλες, Σομαλία, στο Τζιμπούτι, στην κένια κτλ. Όλοι αυτοί βοηθούν την παροχή πληροφοριών προς τους εισαγγελές αλλά και τα θέματα επιμελητίας. Όπως είπαν και οι τελευταίοι ομιλητές, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση στοιχείων. Η Αταλάντα έχει ένα τέτοιο σύστημα και στο Northwood που είναι το στρατηγείο της, αλλά και μεταξύ των ε, αξιωματικών συνδέσμων και στα πλοία υπάρχει ένα δίκτυο της Αταλάντα το οποίο μπορεί να διαβιβάζει πληροφορίε σε εμπιστευτικό επίπεδο και βοηθάει πάρα πολύ τη ροή πληροφοριών. Τέτοιου είδου συστήματα μα επιτρέπουν να έχουμε επιτυχή δίωξη και δίκη των ενόχων. Τι έχουν από κοινού η Αταλάντα και η Σοφία. Έχουν από κοινού το γεγονός ότι η διακινητές που συλλέγονται στη Μεσόγειο και οι πειρατές που συλλαμβάνονται στον Ινδικό δεν είναι οι αρχηγοί των δικτύων, είναι οι απλοί φαντάροι κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι τα εκτελεστικά στοιχεία. Δεν υπάρχει πραγματική συνεργασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους αρχηγούς. Βοήθεια των κρατών δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λέει και η κυρία Φώτη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν λοιπόν τα πρώτα σχόλια των μελών του πάνελ. Πάρα πολύ. πλοκό είναι αυτό το θέμα. Όλοι μας ίσως έχουμε εντυπωσιαστεί από το εύρος των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν θα θέλαμε να υπάρξει εθιμορρησία των υπευθύνων για εγκλήματα διακίνησης ανθρώπων, η πειρατεία. Και όμως είναι τόσο πολύπλοκα τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την δίωξη αυτών των ανθρώπων, όχι μοναχά σε σχέση με την κρίση της ε, μετανάστευσης. Βλέπουμε να υπάρχουν οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις πίσω από όλα αυτά με διασυνδέσεις σε ήδη υπάρχουσες ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τα μέλη του πάνελ και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση γνωρίζουν ότι κάπως έχουν καταπονηθεί τα μέλη των επιτροπών μας μετά από το τόσο ενδιαφέρον πρώτο πάνελ. Ίσως ο κύριος Έλλας θα ήθελε να παρέμβει εδώ και να ξεκινήσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σκάλια, τον κύριο Μάιερ Κάμπρι και τον κύριο Σίλβια για την έλευσή του εδώ. Νομίζω για να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση της, ε, των δικών μας προθέσεων θέλουμε να τονίσουμε και τη σημασία του έργου τους. Έχουμε φυσικά ως Κοινοβούλιο το δικαίωμα εποπτείας και είμαστε υπεύθυνοι και για τη δημιουργία του καταλλήλου πλαισίου και φυσικά έχουμε και αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού. Ένα όμως από τα αντικείμενα αυτής της ακρόασης να σας ευχαριστήσουμε για το έργο σας. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξή. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματική μορφή της οργανωμένης διακίνησης. Μιλάμε πολλές φορές στη διαδικασία αυτή της διακίνησης ως παραβίαση του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά η διάσταση αυτής της οργάνωσης των διακινητών καταδεικνύει ότι υπάρχει και ένα συναφές θέμα που είναι η διαφθορά. Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να τεκμηριώσουν την διάσταση των προβλημάτων διαφθοράς. Πολλές φορές αυτή η διαφθορά Ε, συνδέεται με καταστάσεις που συνδέονται με, την, με το ταξίδι των ε, μεταναστών μπορεί να είναι παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα μπορεί να υπάρχουν λοιπόν πολλές πτυχές διαφθοράς και παραποίησης που συνδέονται με αυτή τη διακίνηση. Για μένα όλα αυτά έχουν μια σαφή διάσταση, είναι φυσικά το παράνομο του στοιχείο και δεύτερον είναι μια προβληματική κατάσταση για τις χώρες αυτές. Βλέπετε σε χώρες των Βαλκανίων χάρη ότι υπάρχει ενδημική διαφθορά ακόμα και οι αστυνομικέ δυνάμεις ε, παίζουν ρόλο στην, ε, αντιμετω... στην διευκόλυνση των, των, της διακίνησης των μεταναστών. Βλέπουμε λοιπόν και κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε πολλές κοινωνίες της Αφρικής. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό θέλουμε εμεί να αντιμετωπίσουμε ή τουλάχιστον να τεκμηριώσουμε αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς. Δεύτερον, κάτι που και αυτό συνδέεται σε αυτό το θέμα είναι το ζήτημα στις ε, χρήσεις συστηματικής βίας έναντι των ε, μεταναστών. Ξέρουμε ότι υπάρχει διαδικασία συστηματικού βιασμού. Πολλές φορές υπάρχει συστηματική χρήση βίας εναντίον τους στα διάφορα στάδια του ταξιδιού. Υπάρχει η τάση να χρησιμοποιούνται για καταναγκαστική εργασία, χάνουν τα χρήματά τους, μετά τους υποχρεώνουν να δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν το ταξίδι τους και δεν ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Μερικές φορές μπορεί να πρέπει να κάνουν καταναγκαστικά έργα για χρόνια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο. Χρειαστήκαμε κάποια χρόνια να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της πειρατείας, αλλά το θέμα τι γίνεται με τη διακίνηση. Όλα αυτά δεν είναι αδίκημα κατά του εθνικού δικαίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ίσως δεν θα υπάρξει δίωξη από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από τις χώρες πρόλευσης, γιατί δεν τους απασχολεί αυτή. Αλλά κάποιος δεν πρέπει να κάνει τη δίωξη αυτή. Υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη διαπίστωση ότι υπάρχει μια διεθνής ε, διάσταση στην ανάγκη να τεκμηριώνονται όλες αυτές οι ενέργειες και αν πρέπει και να υπάρξει και μια δίωξη σε διεθνές επίπεδο. Χρειαζόστε λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση για τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά που έχουν συλλεγεί ως τεκμηρίωση έχουν υποστηριχθεί από τον Διεθνή Οργανισμό για το Έγκλημα και τα Ναρκωτικά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμβάλει ιδιαίτερα. Ποια είναι λοιπόν η διεθνής διάσταση στο επίπεδο της τεκμηρίωσης και πέραν αυτού, κατανοώ ότι έχετε να αντιμετωπίσετε τεράστιες προκλήσεις μόνο και μόνο να αντιμετωπίσετε το θέμα και μόνο της ε, διακίνησης. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα προβλήματά σας, αλλά και η ευρύτερη διάσταση δεν πρέπει να παραμεληθεί, γιατί και η διαφθορά είναι κομμάτι του προβλήματος και μπορεί να οδηγήσει και σε πιο αντικές συνέπειες στο μέλλον, επέκεινα της ε, προσωπικής ε, περίπτωσης ενός αξιωματούχου ενός θεσμού που την χάνει διαφθοράς. Ευχαριστούμε η κυρία Λαριστίν της Λίμπε. Ε, thank you very much and thank you very much for organizing this. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών αλλά παρεμφερών ε, καταστάσεων και νομικών πλαισίων και θεσμικών πλαισίων όπως είναι η λαθρέα διακίνηση και η πειρατεία. Η ερώτησή μου στρεφτεί προς την Eurojust. Τι μπορεί να μάθει κανείς και τι μπορεί να κάνει ώστε να διασφαλιστεί ότι η καταπολέμηση της λαθρείας διακίνησης θα γίνει τόσο αποτελεσματικά όσο είδαμε ότι έγινε και με την πειρατεία. Και η άλλη μου ερώτηση, επειδή εδώ είδαμε συγκεκριμένα νούμερα για τις ε, αποτελεσματικές διώξεις, τι μπορείτε να μας πείτε για τη λαθρέα διακίνηση πόσες υποθέσεις, τι ποσοστό του δικτύου διακίνησης έχει συλληφθεί και διωχθεί. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια, κάποιες ερωτήσεις ε, προς και τους τρεις ε, ομιλητές του πάνελ. Επειδή η λαθρέα διακίνηση ανθρώπων μέχρι τώρα ενέπτε στις αρμοδιότητες της Frontex περισσότερο. Διότι έχουν και την τεχνογνωσία για το θέμα αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, υπάρχει τρόπος ε, να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση στον τομέα της δίωξης και να το χρησιμοποιήσουμε για τη δίωξη των λαθρέων διακινητών μεταναστών. Δεύτερον, ε, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο όρος ε, επιχειρηματικό μοντέλο των ε, διακινητών. Πρόκειται για, ένα, για αποτρόπαια εγκλήματα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Εσείς λοιπόν Τι άλλους τρόπους μπορείτε να σκεφτείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν όλοι αυτοί για το ξεπλήμα χρήματος. Και πώς θα αναγνωριστεί αυτό σε εγκληματική δραστηριότητα των χερσαίων ομάδων. Στις αποστολές μας στο Τουράμ ε, ουσιαστικά ήδη συζητούσαμε τα αποτελέσματα των τρεχουσών ε, επιχειρήσεων της UNAFOR Σόφια και στο πλαίσιο του μηχανισμού SAID και πολλές χώρες συνέβαλαν ε, στην οικοδόμηση αυτών των για αυτό το θέμα του legal finish ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Εδώ ολοκληρώνεται η ερωτήση νομίζω, σωστά. Μάριο Κιούρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια σύντομη αλλά σημαντική ερώτηση. Ε, για τα όσα είπε ο κύριος Δησίλβα στο κέρας της Αφρικής έχουμε καταφέρει να βρούμε εταίρους δεν κάποια ευρωπαϊκά κράτη εκεί μας ε, βρήκαν εταίρους ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε διώξη τους εγκληματίες γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στη λεκάνη της Μεσογείου οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνονται προς τα κράτη της Ευρώπης. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία από τους ίδιους τους μετανάστες γνωρίζουμε τις προθέσεις των διοργανωτών ε, της λαθρείας διακίνησης γιατί δεν μπορούν να διωχθούν ε, στη χώρα τα σύνορα της οποίας προσπάθησαν να περάσουν παράνομα. Εάν υπάρχουν νομικές αιτίες που το εμποδίζουν αυτό, τι είδου μέσα θα μπορούσαμε να ε, δημιουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να τους θέσουμε πρώτον ευθυνοτούς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στους ομιλητές του πάνελ, ξεκινώντα από τον εισαγγελέα τον κύριο Σκάλια. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε μπορείτε να αναλύσετε και ζητήματα που τέθηκαν προηγουμένως. Θα χωρίσουμε τώρα το χρόνο χοντρικά στους στα τρία μέλη του πάνελ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη ερώτηση σχετιζόταν με τη διαφθορά νομίζω. εμείς έχουμε επιληθεύσει την ύπαρξη διαφθοράς στη Λιβύη. με επιπληρωμή ε, διαφεύγουν από τις λιβικές φυλακές ε, οι μετανάστες. Το γνωρίζουμε από τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Αυτό μας διαβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι για τους διακινητές οι μετανάστες είναι οικονομικό αγαθό, όχι ανθρώπινα όντα. Ε, σίγουρα υπάρχει και διαφθορά όσον αφορά την παραποίηση αδειών εργασίας, αδειών διαμονής και αυτή τη στιγμή τρέχουν έρευνες μάλιστα και για ένα δίκτυο λευκών γάμων που πραγματοποιούνται στην Ιταλία με υπηκόους ε, τρίτων χωρών ε, ε, και ειδικότερα από χώρες της υποσαχαρίας Αφρικής ώστε οι πολίτες αυτών των χωρών να μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη ως συνάπτοντες λευκούς γάμους και κάτι άλλο πολυθεύει και αφορά την Ιγυρία συχνά το ταξίδι καταβάλλεται όσον αφορά τις γυναίκες μέσω της πορνείας. Εσείς με ρωτήσετε τι μπορούμε να κάνουμε. Στο πλαίσιο των διαδικασιών μας βοηθάει η συνθήκη του ΟΗΕ του 2000 που προβλέπει όταν υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση οι δραστηριότητες τις οποίες ε, λαμβάνουν χώρα και στην χώρα που πραγματοποιεί την έρευνα τότε μπορεί να προχωρήσει κανείς μπορεί να ασχίσει δίωξη. Ωστόσο αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά και τις άλλε ερωτήσει που έγιναν στη συνέχεια. Για να διώξει κανεί κάποιον για πράξεις ξεπλήματο ε, ξεπλήματος μαύρου χρήματος ή διαφθοράς όταν έχουν διαπραχθεί εν μέρη στο εξωτερικό και ολοκληρώνονται στις ευρωπαϊκές χώρες ή στην Ιταλία, ε, τότε υπάρχει δυνατότητα Όταν όμως δεν έχει συνέπειες στις δικές μας χώρες, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν νομικές δυσκολίες. Διότι εμείς με πολλές από τις χώρες αυτές δεν έχουμε κάποια συμφωνία απέλασης ούτε διεθνείς συνθήκες. Οπότε, όπως είπα προηγουμένως, αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες για να προβούμε στη σύλληψη, όχι στην ταυτοποίηση, αλλά στη σύλληψη ορισμένων από του μεγάλου διακινητέ. Φανταστείτε ότι εμεί, ακόμη και για τι πολύ ε, σοβαρέ ποινέ που έχουν επαγγείλει τα δικαστήριά μα, είχαμε μια πρώτη υπόθεση συνεργασία ε, από έναν από του μετανάστε που καταδικάστηκε, αλλά οι δηλώσει του οποίου και που κατηγορούσαν ε, διακινητές απορρίφθηκαν Εάν ε, είχαμε περισσότερες τέτοιες καταδίκες, ε, θα μπορούσαμε να εξοπλίσουμε και αυτά τα υποφελή στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση, ε, να πω κάτι να δώσω το λόγο στον Γερμανό συνάδελφο για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να παρέμβω, διότι αναφέρατε τρίτες χώρες. Αλλά, για παράδειγμα, οι τουρκικές δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν διεξάγει έρευνα σχετικά με το προφίλ των διακινητών και υπήρχαν σαφή στοιχεία δωροδοκίας αστυνομικών στα Βαλκάνια. Μιλάμε για κράτη-μέλη κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εντός της Μεσογείου, ναι, μπορεί να έχετε δίκιο όσον αφορά την Ιγυρία ή, της, ή τη Δυτική Σαχάρα, αλλά χώρες κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ή και υπό διαδικασία προσχώρησης είναι πιο προσιτή σε έναν εισαγγελέα από την Ιταλία ή την Eurojust. Κύριε Σκάλια, θα θέλατε να απαντήσετε σε αυτό. Εκτός μικροφώνου ο κύριος ομιλητής. Ακούγεται. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό δεν εμπίπτει στις δικές μου αρμοδιότητες, είτε δικαστικές είτε προσωπικές, γιατί εμείς δεν ασχολούμαστε με εγκλήματα τα οποία διαπράττονται σε άλλα κράτη και που δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στη δική μας επικράτεια. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μάλλον πολιτικό πρόβλημα, παρότι ε, καταρχήν είναι δικαστικό. Είναι πολιτικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να βρει τα μέσα και τα εργαλεία για να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Εδώ μιλάμε για άγνωστα εδάφη. στο... Αναφερθήκατε στο θέμα της μετάφρασης. Δεν έχουμε εμπειρία όπως ε, με την διακίνηση ναρκωτικών ε, όπου έχουμε εμπειρία. Ο συνάδελφος της Eurojust πριν λίγο είπε ότι χρήσιμο θα ήταν να βρούμε κάποιες ε, επιχορηγήσεις για τις μεταφράσεις. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ομιλούν διαλέκτους πολυπίκυλες και ακατανόητες. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Χθε μου τηλεφώνησε ένα άλλος από το Παλέρμο, είχε λάβει μου χαρά μια σύλληψη και σύμφωνα με τον κανονισμό μας ε, οι κατηγορίες, ε, τα σχετικά έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν και εμεί αναγκαστήκαμε να βρούμε έναν μεταφραστή ο οποίο μα είπε ναι μπορώ να σα το μεταφράσω αλλά να έχετε υπόψη σας ότι η δική μας διάλεκτος είναι προφορική, δεν υπάρχει γραπτή διάλεκτος οπότε χρειάστηκε να βρούμε, να επινοήσουμε μια λύση ουσιαστικά να μαγνητοφωνήσουμε τις κατηγορίες και να, να τις βάλουμε να τις ακούσει ο κατηγορόμενος. Δηλαδή μερικές φορές τα προβλήματα υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ε, και πολιτικό το πρόβλημα και ειδικότερα με την Τουρκία, κατά την άποψή μου. Κύριε Κλάσμα Κάμπρι, ευχαριστώ πολύ και εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά τα ερωτήματα που τέθηκαν. Η Eurojust αντιμετωπίζει το θέμα της παράνομης διακίνησης μεταναστών όχι μόνο την ε, διέλευση των συνόρων, αλλά το ευρύτερο πλαίσιο. Η διαφθορά φυσικά διαδραματίζει ένα τεράστιο ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε εμπειρία στον τομέα αυτό και το ίδιο ισχύει για τη λαθεμπορία ανθρωπίνων όντων. Δεν είναι μόνο το θέμα της ε, ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή της εργασιακής εκμετάλλευσης. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν σχήματα τα οποία επαναλαμβάνονται στο χρόνο και στο χώρο. Πολλές φορές η διακινητές είναι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι στο παρελθόν είχαν εμπλακεί στην λαθρεμπορία ανθρώπινων όντων για σεξουαλική ή άλλη εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που έχει αποκτήσει η Eurojust στο θέμα της ε, λαθρεμπορίας ανθρώπων στην περίπτωση της ε, παράνομης διακίνησης μεταναστών. Όπως όμως είπε και ο Ιταλός ε, συνάδελφος, ο εισαγγελέα ο, ο οποίος αντιμετωπίζει τέτοια θέματα έχει κάποια εργαλεία ήδη με την προηγούμενη πείρα να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Το θέμα τη διαφθορά είναι πολύ σημαντικό σε όλα αυτά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί είμαστε απλώ μια κοινή λέσχη, υπάρχει ο θεσμικό ιστό, η θεσμική αυτή διαδικασία εμπιστοσύνη. Όταν συνεργαζόμαστε με τρίτε χώρες εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Eurojust προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με κάπως πολλές φορές διαφορετικό τρόπο. Η Επιτροπή ΛΥΠΕ ενέκρινε συμφωνίες συνεργασία με την Ουκρανία, με το Μαυροβούνιο, με την ε, ε, πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προσπαθούμε έτσι να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη που προχωρήσουμε σε τέτοιες συμφορίες και να τις υλοποιήσουμε, πρέπει να δούμε ότι θα τηρηθεί και το κράτος δικαίου. Αυτό αφορά και θέματα προστασία δεδομένων. Υπάρχουν χώρες οι οποίες προχωρούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει θέληση να το κάνουν αυτό. Στην περίπτωση άλλων τρίτων χωρών τα πράγματα είναι πιο πεπλεγμένα. Αν δεν έχετε μια κυβέρνηση με την οποία να διαπραγματευτείτε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν δεν έχετε, έχετε όλα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου να αντιμετωπίσετε με τις χώρες της Μέσης Αντώνης και της Βόρειας Αφρικής, προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε ένα διάλογο, να έχουμε σημεία επαφής, ώστε αν θέλετε να στείλετε μια επιστολή να ζητήσετε πληροφορίες, τουλάχιστον Έχετε κάποιον στον οποίο να στείλετε αυτά τα στοιχεία για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτά είναι απλώς μια αρχή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία του να οριστικοποιήσουμε αυτό το οποίο προβλέπει και η οδηγία του Eurojust, να υπάρχουν ε, εισαγγελείς ε, σύνδεσμοι και το επόμενο ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα αποτελεσματικά. Και πάλι είναι θέμα χρηματοδότησης, αφαιρών. Χρειάζεται να στείλετε κάποιον σε μία από τις χώρες αυτές της ε, Μέσα Ανατολής Βόρειας Αφρικής. Πρέπει να είναι κάποιος εισαγγελέα ο οποίος ξέρει τη γλώσσα και τα τοπικά έθιμα. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας για τα άτομα αυτά. Χρειάζεται χρηματοδότηση. Προτού κάποιος τέτοιος ε, σύνδεσμος είναι λειτουργικός, χρειάζεται και μία συμφωνία με την αντίστοιχη χώρα, ώστε να υπάρχει και ένα πλαίσιο με στο οποίο μπορεί να εργαστεί ο εισαγγελέα αυτός. Και στη συνέχεια πώς θα κάνετε το ένα ή το άλλο, Ενδεχομένω θα έχετε κάποιους ε, διακινούμενους συνδέσμους ή κάποιους οι οποίοι είναι μόνιμοι εκεί. Υπάρχει εκεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από τον Γάλλο σύνδεσμο εισαγγελέα στην Τουρκία που μας έδωσε πολλά στοιχεία σε σχέση με το πώ λειτουργεί το σύστημα αυτό και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε λειτουργικό το σύστημα αυτό και να τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Και όπως είπα στην αρχή, αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια ουσιαστική διαδικασία δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή είναι μεγάλη κρίση μπορούμε να παραλείψουμε κάποια στοιχεία της ένδικης διαδικασίας. Δεν μπορούμε να δικάζουμε άτομα χωρίς τη σωστή διαδικασία, χωρίς μετάφραση, χωρίς σεβασμό των δικονομικών κανόνων. Όλα αυτά τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για να γίνει σεβαστό και το δικαίωμα της υπεράσπισης για τον οποιοδήποτε κατηγορούμενο και ένα στοιχείο που αναφέρατε και το οποίο είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τη Eurojust και εργαζόμαστε για το θέμα αυτό πάρα πολύ εντατικά. Το θέμα είναι το θέμα της κατάσχεσης στοιχείων ενεργητικού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν διακινούν μετανάστες επειδή έχουν καλή ψυχή ή για την ψυχή της μητέρας τους, αλλά διότι θέλουν να μαζέψουν χρήματα. μπαλιόκο. Είναι λοιπόν πολύ πιο δύσκολο να μπορέσετε να κατασχέσετε τα στοιχεία του ενεργητικού τους γιατί ουσιαστικά είναι ρευστό χρήμα αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν και αποκτούν από αυτές τις ενέργειες. Για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει κάποια δίωξη, θα πρέπει κάποιος να αποδείξει γιατί έχει τα στοιχεία αυτά, να έχει ένα απόθεν έσχες βέβαια. Μονάχα στις περιπτώσεις που είναι συντριπτικά τα στοιχεία μπορεί κανείς να αποδείξει κάτι. Στις άλλες όχι. Προσπαθούμε λοιπόν να πληροφορήσουμε τους ε, ομολόγους μας αν θέλουμε να κάνουμε μια κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού να ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα σε πρακτικό επίπεδο που πρέπει να αντιμετωπίσουν και αυτά πρέπει να γυρίσουν μετά στον νομοθέτη, να πούμε να τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε πολλές περιπτώσεις, ίσως θέλετε να τροποποιήσετε την νομοθεσία ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Στο προηγούμενο αξίωμά μου είχα πολλές συναντήσεις και συζητήσεις με τους Ιταλούς νομοθέτες γιατί πολλές φορές η κατάσταση στη χώρα μου δεν ήταν αυτή που περιμένανε να είναι οι Ιταλοί συνάδελφοί μας. Αλλά πρέπει να βρείτε έναν τρόπο συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εναρμονισμένο ποινικό δίκαιο, απλώς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε την ύπαρξη συνόρων στην Ευρώπη. Αυτά κάνει η Eurojust δεν είμαστε τόσο ανόητοι που να πιστεύουμε ότι ο κόσμο τελειώνει στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα και με τρίτε χώρε, βήμα-βήμα. Έχουμε κάνει προσπάθειε συνεργασία σε μεγάλε τρομοκρατικέ υποθέσει, όπου είχαμε συναδέλφου από την Τινησία που συνεργάστηκαν μαζί μα. Ο κόσμο δεν είναι βέβαια μαύρο ή άσπρο, δεν είναι μοναχά οι καλοί και οι κακοί. Πρέπει να βρούμε εταίρου σε ορισμένε περιπτώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ζητήσατε στατιστικά στοιχεία πόσες ε, υποθέσεις έχουν εκδικαστεί. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα να σας το πω γιατί ο ρόλος μας στη Eurojust είναι να διευκολύνουμε την συνεργασία των εισαγγελέων και των δικαστηρίων. Να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν στην απαγγελία κατηγορίας όταν χωρί λόγος αλλά δεν παίρνουμε όλες τις πληροφορίες από αυτούς για το ποια ήταν η τελική απόλυψη της δικαστικής διαδικασίας. Προσπαθούμε τουλάχιστον, ιδίω σε περιπτώσεις δικών για τρομοκρατικά δικήματα, να συλλέξουμε στοιχεία και να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω ο κ. Κόνιξ είχε δώσει μια αναφορά στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για τα θέματα αυτά. Για τις περιπτώσεις όμως μετανάστευσης, είναι ακόμα ένα καινούριο πρόβλημα. Αυτό το οποίο είδα είναι μια αύξηση της ανάγκης για περισσότερο συντονισμό και συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια. Προηγουμένως ήταν έτσι και έτσι τα πράγματα, δεν ήταν τεράστια ανάγκη, τώρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αυτή η ανάγκη και δεν είμαστε τόσο προχωρημένοι που να μπορούμε να πούμε να αυτό το ποσοστό περιπτώσεων έχει παραπευθεί στο δικαστήριο. Ο κύριος Τεσίλου τόνισε πόσο χρόνο μπορεί να παίρνει μια διαδικασία και αυτό εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προβλήματος και κάτι ακόμα που είναι πολύ δύσκολο και το είπε και ο κύριος Τεσίλου προηγουμένως είναι ότι πολύ συχνά πιάνετε πρώτα τα μικρά ψάρια. Στην περίπτωση αυτή του φορτηγού με τους 71 ε, μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους πιάσαν τους δύο οδηγού, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι πίσω από αυτούς και αυτούς θέλουμε να πιάσουμε. Και αυτό χρειάζεται χρόνο και πολλή προσπάθεια. Χωρίς συντονισμό όμω, χωρίς συνεργασία, ποτέ δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. the... Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ντεσίλβα, θα ήθελα να κάνω μια επιπλέον ερώτηση. η οποία σε κάποιο βαθμό σχετίζεται με τις προηγούμενες παρατηρήσεις ε, του κυρίου Μέιερ Πέμπρη. Κατά την επίσκεψη της ΣΕΝΤΕ στα αρχηγείο της Αταλάντα κάναμε μια σύντομη συζήτηση για πιθανές ε, σχέσεις μεταξύ των εγκλήματων πειρατείας με ορισμένες τρομοκρατικές ομάδες ε, στο κέρας της Αφρικής. Επίσης, ε, από τα σημερινά σημεία στην ημερήσια διαταξή της ΣΕΝΤΕ, μάθαμε για την ε, αυξανόμενη επιρροή του Ισλαμικού κράτους στη Λιβύη. Πιστεύετε ότι υπάρχουν παρόμοιες σχέσεις με τις αλυσίδες ε, λαθρέας διακίνησης μεταναστών και ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σχέσεις τέτοιες με τα τρομοκρατικά δίκτυα, ε, χρηματοδότηση των τρομοκρατών μέσω τέτοιου είδους δραστηριοτήτων επίση. Πρέπει να πω, δεν ε, έχω αρμοδιότητα για να σας πω κατά πόσο έχουν αποκαλυφθεί τέτοιες σχέσεις ε, από το Σοφία μεταξύ τρομοκρατικών ενεργειών και λαθρείας διακίνησης. Το, η επιχείρηση Αταλάντα είχε δώσει κάποιες ενδείξεις αλλά δεν, υπάρχει, δεν έχει διαπιστωθεί η σχέση. Για να απαντήσω σε κάποια από τα άλλα σημεία τα οποία τέθηκαν. Ε, πρώτα απ' όλα η κατάσχεση περισσοκών στοιχείων η επιχείρηση Αταλάντα επιτρέπεται να κατασχέσει ε, περιουσιακά στοιχεία σωμαλών πειρατών ε, δύναμη του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και μέσω της ανταλλαγής επιστολών που δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τις περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε απαραίτητα να αποδείξουμε ότι κάποιος ε, έχει διαπράξει πειρατεία αλλά για εύλογους λόγους πιστεύουμε ότι το έχει κάνει μπορούμε να, παρόλα αυτά να κατασχέσουμε τα περιουσιακά τους ε, στοιχεία χωρίς να τους πάμε στα δικαστήρια. Αν βρούμε δηλαδή ένα σωμα... πλοίο με σημαία Σομαλίας ε, και δεν έχουν όπλα, αλλά, έχουν πολύ αλλά αυτό το πλοίο έχει πολύ ισχυρού κινητήρε. Ε, οι άλλα στοιχεία που μα αποδεικνύουν ότι μπορεί να διαπράττει πειρατεία μπορούμε να το κατασχέσουμε. Αν βρούμε ένα φουσκωτό με λιγότερο δυνατό κινητήρα, Ε, ε, και του βάλουμε σε ένα φουσκωτό δηλαδή, για να του στείλουμε πίσω στι ακτέ τη Ομαλική ακτή και κατασχέσουμε το πλοίο ώστε να του αφαιρέσουμε δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο στο μέλλον. Για την εναρμόνιση του ποινικού συστήματο ε, αυτό είναι αδύνατο και με την πειρατεία. Για παραδείγμα, η μικρότερη ποινή που έχω δει πρόσφατα σε ένα δικαστήριο των Σεχελών ήταν τρία έτη. Το ρεκόρ ήταν 439 ημέρες από ένα ισπανικό δικαστήριο αλλά το, η μέγιστη ε, ποινή στην Ισπανία είναι ουσιαστικά 30 χρόνια. Όλα εξαρτώνται από το πώς θα αντιμετωπιστεί κανείς. Ε, οι ανήλικοι 118 ε, δικάζονται από τοπικά ε, συστήματα όσον αφορά την ποινή τους. Οι Σομαλοί πειρατές που έχουν συλληφθεί από τα Ταλάντα δεν είναι ανόητοι έχουν παρατηρήσει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις οι ανήλικοι ε, καταδικάζονται για τρία χρόνια και οι ενήλικες για 14 οπότε τώρα λένε όλοι ότι είναι ανήλικοι. Οπότε, ξέρετε, μετά χρειάζεται επιπλέον κόστος για το Αταλάντα ώστε να φέρει ειδικού που μπορούν να αποδείξουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ενήλικες. Όλα αυτά λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμεί στο κέρα Αφρική θα τα ζήσετε και στην Λιβύη. Κανένα δεν πρόκειται να προσπαθήσει να αποδείξει την ηλικία του με ένα προσωπικό γέννη. Θα σα πούν τι ηλικία έχουν και μετά θα απαιτήσουν την αναλογία αντιμετώπιση. Τώρα, όσον αφορά τα νομικά εργαλεία που χρειαζόμαστε, όπω είπε και ο συνάδελφο ο κ. Μάια Κάμπρη, τρία νομικά εμπόδια χρειάζεται να ξεπεράσουμε για να μπορέσουμε ε, Πρώτα χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση με την οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Στι Σεχέλε, στο Μαυρίκαιο έχουμε δημοκρατικέ κυβερνήσει που λειτουργούν και με τι οποίε μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Επίση, χρειαζόμαστε ένα εθνοοικονομικό σύστημα που να μπορούμε, στο οποίο να μπορούμε να βασιστούμε. Η πειρατεία, όπω ανέφερα προηγουμένω, αποτελεί παγκόσμιο αδίκημα ο ορισμός της πειρατείας ε, βρίσκεται στη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τους νόμους της θάλασσας. Αλλά δεν μπορεί κανείς να βασιστεί μόνο σε αυτόν τον ορισμό για να πει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Χρειάζεται εθνική εγχώρια νομοθεσία που να την καθιστά παράνομη και να ε, προβλέπει συγκεκριμένες ποινές και σε κάθε χώρα αυτό πραγματοποιείται διαφορετικά. Πρόσφατα έχουμε δει ότι ορισμένε χώρε έχουν πάρει τον ορισμό από τη συνθήκη των ΗΠΑ και την έχουν αντιγράψει επακριβώ στου εθνικού νομικού κώδικε. Στο παρελθόν υπήρχαν μικροαλλαγέ, οπότε έπρεπε να αποδείξει κανεί διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τη δικαιοδοσία που χρησιμοποιούσε. Όπω είπα λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχει μια εθνική νομοθεσία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Σομαλία, διότι η Σομαλία δεν αναγνωρίζει ως έγκλημα την πειρατεία ομοσπονδιακά ε, αφού δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ε, ως ομοσπονδιακό κράτος η Σομαλία δεν αναγνωρίζει την πειρατεία ως έγκλημα δεν μπορεί δηλαδή να πάει κανείς να διώξει κάποιον σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μογκαντέσου αφού υπάρχει λοιπόν ένα κράτος και μια εθνική νομοθεσία πρέπει να μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, της Εθνικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή, κατά πόσο δεν θα, θα είναι ασφαλής κάποιος, ε, δεν θα, δεν θα υποστεί βασανιστήρια ή την θανατική ποινή. Δεν μπορεί δηλαδή να απελάσει κάποιον στην Εμένη όπου υπάρχει θανατική ποινή, ούτε στην Ινδία, γιατί και στην Ινδία η πειρατεία τιμωρείται με θανατική ποινή. Χρειάζεται λοιπόν μια εθνική νομοθεσία Χρειάζεται να υπάρχει σεβασμό προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια κυβέρνηση με την οποία κανεί να μπορεί να διαπραγματευτεί. Τώρα, στο πλαίσιο τη επιχείρηση Αταλάντα, ε, συζητήσαμε την επικαιροποίηση των εθνικών νομοθεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, ο Μαυρίκιο πήρε τον ορισμό τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τη θάλασσα την αντέγραψε στη δική τους θαλάσσια πράξη για τη, ε, στην πράξη για τη θαλασσία και την πειρατεία αλλά έχει ένα σύστημα αποδεικτικών στοιχείων που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η βεντοδιάσκεψη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο, κάποιος κάποιον μέσα σε ε, μια αίθουσα ανάκριση. Ε, δεν ξέρω το σύστημα αυτό υπάρχει και στην Ιταλία. Αυτοί είναι οι τρει παράγοντε πάντω. Είναι η, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια κυβέρνηση με την οποία μπορεί κανεί να διαπραγματευτεί και μια εθνική νομοθεσία. Well, gentlemen. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές και από τα δύο πάνελ. Ήταν πολύ τεχνική η σημερινή συζήτηση. παρόλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας αύριο το πρωί στις 9. Σας ευχαριστώ.